Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να ξεκινήσουμε ε, διότι δεν πρέπει να παίρνουμε κακές ε, συνήθειες αλλά ξέρετε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος είμαστε μεταξύ τριλό, τριμερούς διαλόγου και ε, συνδιαλλαγής και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε και προτείνω να ξεκινήσουμε. Έχετε καταρχήν την ημερήσια διάταξη μπροστά σας και προτείνω μερικές ε, αλλαγέ σχετικά με τα σημεία 13 και 14 κατόπιν ετήσεω του εισηγητή κυρίου Γκοτμάνη αποσύρονται το σημείο 5 είναι πολύ σημαντικό και θα το εξετάσουμε αμέσως μετά από τις ανακοινώσεις του Προέδρου και ε, την παρουσία του Επιτρόπου Λεβαντόφσκη ο οποίος θα έρθει να μας παρουσιάσει ε, τα, τις απόψεις του το οποίο έχει κάνει εντάχει στην τελευταία ολομέλεια και θα μπορέσει τώρα να μας δώσει ορισμένες διευκρινήσεις και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής στο στάδιο αυτό καθότι όλα αυτά είναι σημαντικά για την διαπραγμάτευση του προπολογισμού του 2011. Σχετικά με τον προπολογισμό του 2011 έχουμε ε, προβλέψει σήμερα το απόγευμα και κλεισμένων των θυρών. Μεταξύ μας δηλαδή 3 με 4 μία συζήτηση εδώ και ε, το διευκρινίζω για τις προσωπικότητες που ενδιαφέρονται για τις ε, εργασίες μας ότι 3 και 4 το απόγευμα σήμερα θα συνεδριάσουμε και κλεισμένων των των Τα σημεία 6 και 7, δηλαδή ε, την πολιτική των ε, κτηρίων και τον ε, προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα τα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, την παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Σας καλωσορίζω μόλις ξεκινήσαμε και υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη. Τα σημεία 26 και 27 θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα παρουσία του κυρίου Κράους Βέμπερ και με ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ζητούν εντάχει να συζητήσουμε ε, μη ε, πληρωμή στο σημείο 53 για να βοηθήσουμε τα άτομα τα οποία επλήγησαν από τις πλημμύρες στο Πακιστάν. Οπότε σας έχω διανύμει ένα σχετικό έγγραφο και θα δούμε μέχρι το βράδυ αν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πρόταση του εισηγητή για ένα ιδίως στο, είναι το έμβασμα 54 με συγχωρείτε 54 λέει ο πρόεδρος οπότε έχουμε πέραν αυτού στην ημερήσια διάταξη ένα θέμα το οποίο θα παρουσιάσει ο εισηγητής Ράιμερ Μπέγκερ, ο οποίος μόλις μπήκε καλά εξοπλισμένος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ΙΤΕΡ και το πακέτο της Λισαβόνας για τις συνολικές δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις. Οπότε σήμερα το απόγευμα οι δύο εισηγητριές μας, η Συντόνια και η Έλγα, θα μας παρουσιάσουν το που βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις και ο θα μας παρουσιάσει ε, το πού βρισκόμαστε σχετικά με το ίτερ και το, τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο της Λισαβόνας. Λοιπόν, όσον αφορά τις ε, γλώσσες ε, μπορείτε να τις βρείτε στο κόμπι News και υπάρχει αναμετάδοση στο διαδίκτυο παρόλο που δεν βλέπω κάτι προφανές και στο σημείο 3 2-3 έχετε ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο κοινή αποστολής με ε, ακόμη μία ε, επιτροπή οπότε δεν θα επανέλθω σε αυτό. Σημείο 3. Ο, με συγχωρείτε, ε, σχετικά με την κοινή επιτροπή, με την επιτροπή Κοντ στην Κροατία ε, υπάρχουν πολύ ανητικές απόψεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και ήθελα να κοιτάξουμε αυτές ε, αυτό το θέμα διότι υπάρχουν πολλά θετικά θέματα που προχωρούν στην Κροατία και θα έπρεπε έπρεπε να αναφερθούν. Ευχαριστώ συνάδελφε και εγώ αυτή την εντύπωση είχα προσωπικά και γι' αυτό εν αντιθέσει με το ότι γράφεται στο Κόμπι News δεν θα διανύουμε σε αυτό το στάδιο την έκθεση. Θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε το κείμενο αυτό κατά τρόπον ώστε το κείμενο το οποίο θα κυκλοφορήσει να αναφέρεται στις απόψεις τις οποίες και εσείς παρουσιάσατε. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Το τρίτο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών της προηγουμένης συνεδρίασης το οποίο μπορούμε να δούμε πολύ γρήγορα γιατί δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 5 και ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι δέχτηκαν τη στιγμή που είμαστε τόσο βεβαρημένοι να παρουσιάσουν την budget review και να τη συζητήσουν μαζί μας. Στην Ολομέλεια παρουσιάστε τις γενικές γραμμές αυτής, αυτού του σχεδίου και που έχουν υποβληθεί και γραπτός. Θα ήθελα τώρα να μας μας υπενθυμίσετε τα βασικά θέματα, τις βασικές καινοτομίες κατά τρόπον ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να αντιδράσουν και ε, να θέσουν ερωτήσεις κατά τρόπον ώστε και εμείς να δούμε ε, πιο σαφώς πού οι προτάσεις αυτές μπορούν ε, να ε, ε, προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό του 11 και για τις δημοσιονομικές προπτικές μέχρι το 2014. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, ε, ειδικά αυτό το μήνα, για συναντήσεις, για ανταλλαγή απόψεων. Ο στόχος μας σήμερα είναι να καταδείξουμε την προσπάθεια που κάνουμε για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία και θα οδηγήσει σε μια νέα ανακοίνωση για το μελλοντικό προϋπολογισμό βάσει της διαδικασίας, της προϊούσας διαδικασίας που βρίσκεται σε κρίσιμη φάση ανάμεσα στον τριμερή διάλογο και στην συνδιαλλαγή. Οι συναρμόδιοι φορείς γνωρίζουν ότι το Κοινοβούλιο θα ήθελε να συνδέσει τα δύο ζητήματα, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με την αναθεώρηση και όχι με την αιτήσια διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού. Η εντολή προς την Επιτροπή ήταν σαφέστατη, αλλά θα έπρεπε να δούμε και για το εισόδημα και για τις δαπάνες, ποιε είναι οι εξελίξεις. Ε, έγινε ευρύτατη δημοιαβούλευση, πάνω από 300 ε, ε, συνεισφορές και μαζί με τον πρόεδρο Λάμα Σουρ συζητούμε κυρίως το ζήτημα των εσόδων Τελικά στη διαδικασία αναθεώρηση του προϋπολογισμού θίξαμε αυτό το ζήτημα και είχαμε διάφορες απαντήσεις από πολλές πλευρές στην Ευρώπη. Ε, είναι ιδιάζουσα η κατάσταση σήμερα. Για πρώτη φορά έχουμε νέες αρμοδιότητες προβλέπονται στη συνθήκη της Λισαβόνας και ταυτόχρονα έχουμε νέες προκλήσεις και ε, ε, ζητούνται κοινέ απαντήσεις. Όχι απαντήσεις από πλευράς των μεμονωμένων κρατών μελών. Αυτό αφενός αφετέρου το κλίμα της αποταμίευσης, της λιτότητας ε, που επικρατεί είναι ε, πιο πρόδειλο από ό,τι ποτέ και επηρεάζει τις εξελίξεις. Τι έπεται το έγγραφο για την συνοχή και για την κοινή ε, γεωργική πολιτική βασικέ, βασικούς τομείς όπου τοποθετούνται οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Σώμα των Επιτρόπων συζητά και το θέμα της διεύρυνσης, το θέμα της Κροατίας, ε, τι είναι θετικό, τι είναι αρνητικό προς την προσχώρηση της Κροατίας, αλλά όχι και μόνο για την Κροατία. Ε, είναι ιδιάζουσα λοιπόν η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Ένα βασικό τμήμα της διαδικασίας αναθεώρησης του προϋπολογισμού έγκυται στην ευθυγράμμιση των αρχών κατάρτισης του υπολογισμού σε αυτό το νέο περιβάλλον και πρέπει να αντλήσουμε επίσης και διδάγματα. Οφείλω να το επαναλάβω, είναι σαφή τα διδάγματα και βλέπω τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο της Λισαβόνας και καταλαβαίνω το βασικό δίδαγμα είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει προβλεψιμότητα όταν ε, οι δικαιούχοι του προϋπολογισμού καλούνται να καταρτήσουν πρόγραμμα, καταλούνται να υλοποιήσουν το προϋπολογισμό. Ε, πληρώνουμε το τίμημα όταν δεν είμαστε παρκώς ευέλικτοι, όταν δεν ε, αντιδρούμε αρκετά γρήγορα. Είναι σαφές το μήνυμα, πρέπει να ορίσουμε το ελάχιστο επίπεδο επίπεδο ευελιξίας. Ε, ποιες είναι οι νέες εξελίξεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη και που δεν είχαμε προβλέψει όταν ναι, εκδόθηκε η εντολή για την αναθεώρηση του προπολογισμού, Τη συνδέεται το ένα και περισσότερο με την οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρώπη, όχι μόνο μέσω των εγγυήσεων, ε, σύναψη δανείου δηλαδή, στον στο μηχανισμό ε, ισολογισμού των πληρώμων, αλλά έχουμε και τον μηχανισμό σταθεροποίηση, ε, που τίνει να παγιωθεί για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και κάτι άλλο που αναμένεται να συμβεί με την πρόοδο των εργασιών ένα toolbox, ένα κυβότιο εργαλείων ε, όχι μόνο ε, για τις υποχρεωτικές καταθέσεις από τις χώρες ε, που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας αλλά και το θέμα των ποινών και του ΔΕΛΕΑΡ που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τον προϋπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις. Τρίτον, ε, το, ε, η μόχλευση που επιζητούμε λόγω των περιορισμών, ε, δηλαδή πρέπει να διευρύνουμε την ικανότητα του κοινού προϋπολογισμού 2,5% των δημοσίων δαπανών και δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως η εθνικοί προπολογισμοί. Πρέπει να διευρύνουμε την ικανότητα μέσα από τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και αυτό είναι το θέμα του τεχνικού παραρτήματος προφανώς. Η ομάδα εργασίας της Επιτροπής ε, κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα και εμεί ε, στην ε, ετήσια αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού για τους καινοτόμου χρηματοδοτικούς μηχανισμούς έχουμε θέσει το ίδιο θέμα και τώρα συζητούνται τα ευρωομόλογα, μια υποδομή για έκδοση ευρωομολόγων ε, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο ε, στην εναρκτήρια ομιλία του όταν έχετε την νέα θητεία ενώπιον του Κοινοβουλίου. Αυτές είναι οι εξελίξεις, αυτά είναι τα διδάγματα. Πώς θα ευθυγραμμιστούμε λοιπόν στο προϋπολογισμό. Δεν έχουμε ε, ακόμη ευελιξία για να προσαρμοστούμε συνθήκε τη Λισαβόνα και στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Αυτό συνιστά μέρο τη ε, προϊούσα διαδικασία. Το έχουμε συζητήσει. Ε, πολλές φορές το θέμα και σήμερα εξάλλου, δηλαδή σε ποιο βαθμό έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε μια τύπου Λισαβόνας αναθεώρηση χωρίς νομική βάση ε, σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις ετήσιες ε, προσαρμογές, ε, όπως γίνεται τώρα δηλαδή αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξ αρχής είναι το τμήμα των ιδίων πόρων προφανώς με έξι υποψηφίους, κανείς δεν είναι τέλειος ε, βέβαια, σε αυτό τον κατάλογο που παρουσιάστηκε με πολλές μελέτες ε, υποβάθρο που έγιναν πριν καταλήξουμε σε αυτόν τον ε, τελικό κατάλογο ανταποκρινόμενοι στα σαφή αιτήματα πολλών πρωτευουσών, δηλαδή δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μειωθούν οι άμεσες εισφορές στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω εξυγίανσης των εθνικών προϋπολογισμών που πρέπει να κάνουν. Βέβαια από τις ίδιες πρωτεύουσες δεν είχαμε επίσημες αντιδράσεις μετά από την υποβολή αυτού του επίσημου αιτήματος, αλλά θα πρέπει να είμαστε και εμείς ανοιχτοί ε, από πλευράς ε, εσόδων. Οι αρμόδιοι για τον προϋπολογισμό ε, που ε, γνώριζαν ότι την Επιτροπή διέρεαν διάφορα ανώνυμα έγγραφα στο παρελθόν. Αυτή τη φορά τίποτα και αποδίδω τα εύσημα σε αυτή την ειδική διαδικασία που εφήρμοσε η Επιτροπή που με αυτονομία ε, ε, διαμόρφωσε για πρώτη φορά κατά αυτόν τον τρόπο την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Κανείς δεν περίμενε το ουσιαστικό περιεχόμενο της πρότασης. Τι διέρεε λοιπόν στο παρελθόν και είναι καλό σημείο αναφορά όταν συζητούμε το περιεχόμενο τη αναθεώρηση του προπολογισμού. Φερρυπίν για τη συνοχή ε, μιλούσαμε για την κεντροποίηση της πολιτικής συνοχής ε, που θεωρείται ως μια αναδιανεμητική πολιτική για τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Τώρα βλέπουμε τελώς διαφορετικά την πολιτική της συνοχής. Ε, θα πρέπει να θεωρήσουμε το ως αναπτυξιακή πολιτική, καλύπτοντας και το θέμα της Δυτικής Ευρώπης των μεγάλων αστικών κέντρων ε, σε επίπε... Ε, ε, μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Δεν επιδιώκουμε πλέον κεντροποίηση της διαδικασίας. Υπάρχει δε μία τάση σε σχέση με το κομμάτι της κοινή γεωργικής πολιτικής στον προϋπολογισμό. Εδώ έχουμε σαφή εξέλιξη, όχι επανάσταση, εξέλιξη Ήμασταν στο 80% τη δεκαετία του 80, τώρα είμαστε στο 40% του προϋπολογισμού ε, και μιλάμε για αύξηση της χρηματοδότησης ε, των φιλοδοξιών της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο μετά ε, την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είναι αδύρυτη ανάγκη να γίνει αυτό και στο κεφάλαιο 1α στο τμήμα 1α μάλλον για τις για το θέμα αυτό, ο στόχος μας είναι να ε, προαγάγουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Δεν προεξοφλούμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ε, ποιες είναι οι αλλακτικές λύσεις, η διάρκεια του δημοσιονομικού ε, πλαισίου, δύο φορές πέντε είπαμε. Τι σημαίνει αυτό. Ε, υποχρεωτική αναθεώρηση στα μέσα οπωσδήποτε και αποθεματικά για ενδεχόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση. Δεύτερον, που είναι επίσης προαιρετικό πώς ακριβώς ε, θα δημιουργήσουμε την δομή του προϋπολογισμού, θα πρέπει να ενοποιηθούν κάποια τμήματα ε, ή να φτιάξουμε τον προϋπολογισμό με βάση τους ε, κυριότερους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Όλα αυτά για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού θα πρέπει να συνυπολογιστούν με τα περιτεχνικού παραρτήματος, διότι Σαλβατόρ ε, Γκαρίγκα ε, είπε ότι δεν μπορούμε βέβαια να βλέπουμε ένα έγγραφο για τον προεκλογισμό χωρί αριθμητικά στοιχεία. Τα αριθμητικά δεδομένα είναι μέσα στο τεχνικό παράρτημα. Πρέπει να τα εξετάζουμε από κοινού. Ε, βέβαια. Γι' αυτό σε διμερεί ανεπίσημε επαφέ έχουμε άπλετε ευκαιρίε να συζητήσουμε το θέμα και σα ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πολλοί ζήτησαν το λόγο και πολλέ. Πρώτος πρώτος ο Σαλβαδόρ Γκαρίγκα που φαντάζομαι ότι θα μιλήσει και ως εισηγητής του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Προπλοκισμών και ως ο ίδιος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω με ποια ακριβώς ιδιότητα πρέπει να μιλήσω τώρα για να απαντήσω σε αυτά που είπε ο Επίτροπος. Έχει μιλήσει και άλλη φορά και στην Επιτροπή Σούρ για την αναθεώρηση του προπολογισμού. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι τον ακούσαμε και τότε μάθαμε πολλά. Καταρχήν λοιπόν πρέπει να διαχωρίσουμε την, το όραμά μας για το μέλλον γενικότερα με τον προϋπολογισμό του 11. Από τον προϋπολογισμό του 11. Ας περιοριστούμε λοιπόν στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού και στα στοιχεία που είχαν τεθεί από την Επιτροπή ΣΟΥΡ. Ο Επίτροπος μας είπε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τη θέση του. Στην προηγούμενη μας συνάντηση λοιπόν είχαμε πει ότι η δομή των επόμενων δημοσιονομικών προϋπολογισμών προοπτικών θα βασιζόταν στη στρατηγική του 2020 και στους τρεις της άξονες, αναπτυξιακούς της άξονες. Είχαμε επίσης πει, όταν κοιτάζαμε τους αριθμούς που μας έδωσε ο Επίτροπος, είχαμε δηλώσει στη Σιδονία ότι τα διάφορα σχέδια ΦΑΡ που είχαν συμπεριληφθεί στον προβλησμό του 2011 δεν ήταν μέρος αναπόσπαστο τμήμα αυτής της στρατηγικής του 2020. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να μας εξηγήσει κάπως καλύτερα ποια είναι η ιδεώδης κατά την άποψή της δομή των νέων δημοσιονομικών προοπτικών που σίγουρα θα είναι πιο απλοποιημένες από τις τωρινές, θα έχουν λιγότερους στόχους αλλά θα είναι πιο συγκεκριμένες όπως λέει στη στρατηγική του 2020 και έπειτα κύριε Επίτροπε αφού θα έχουμε αναλύσει την αναθεώρηση του προπολογισμού και τις προσθήκες αφού το κάναμε μάλλον διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν και πολλά στοιχεία ως προς την απλοποίηση της εκτέλεσης της χρήσης του προϋπολογισμού ενώ είναι κάτι τελείως απαραίτητο αν θέλουμε να βελτιωθεί ο προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια. Μας δώσατε ορισμένες ενδείξεις, είπατε ότι η ικανότητα απορρόφησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών και διοικήσεων για την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων είναι σημαντικός παράγοντας για την επιλεξιμότητα των σχεδίων, ωραία. Αλλά τότε πρέπει και η Κομισιόν να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, να τα δει σε μεγαλύτερο βάθος. Και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το είχαμε πει και τότε, αλλά ας το πω και εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, είναι το εξής. Θέλουμε μέσα στις δημοσιονομικές προοπτικές να συμπεριλαμβάνονται οι στόχοι της στρατηγικής του 2020 που είναι τι, η στρατηγική της Λισαβόνας με προϋπολογισμό. Υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για να γίνει κάτι τέτοιο το μόνο μέσο που διαθέτεται ως Επίτροπος για να διασφαλιστεί το ότι θα εφαρμοστούν πράγματι οι αναπτυξιακοί στόχοι στα εθνικά προγράμματα θα ήταν να το συμπεριλάβετε στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού που προβλέπετε ήδη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αν δεν υπάρξει, δεν δοθεί συνέχεια, δεν παρατηρήσετε πώς ακριβώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα, τότε η στρατηγική του 2020 δεν θα εφαρμοστεί πλήρως και στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές δεν θα θέλαμε να υπάρχουν τέτοιες εγγενείς αδυναμίες. Πρέπει λοιπόν κύριε Επίτροπέ μου να μας το αποσαφηνίσετε, να μας εξηγήσετε καλύτερα πώς ακριβώς έχετε την πρόθεση να συμπεριλάβετε τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε αυτές τις αξιολογήσεις της Κομισιόν. Μάλιστα, παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι, διότι ο Επίτροπος δεν μπορεί να μείνει πάρα πολύ ώρα. Ο James Ellis. Ευχαριστώ πολύ. Τον Επίτροπο για την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να έχουμε κάποιες βασικές ανταλλαγές απόψεων. Η δήλωση του Συμβουλίου της 29 Οκτωβρίου είναι μια βάση που την ξέρουμε και οι δύο πλευρές, αλλά θα ήθελα να πω ότι για μένα είναι πολύ περίεργο να γίνεται ολόκληρη αναθεώρηση του προπολογισμού χωρίς να έχουν αναθεωρηθεί τα ποσά των προγραμμάτων για το 2020 τουλάχιστον από του εθνικά προγράμματα για το 12 και 13. Ήδη χρόνια, δεκαετίες πριν είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση αλλά ούτε τότε είχαν με, αλλάξει οι αριθμοί. Περίεργο αυτό. Δεύτερον, μου φαίνεται επίσης ότι δεν εξηγείται εύκολα το ότι τα προγράμματα πρέπει να αναφέρουν συγκεκριμένα πού διαθέτουν τα χρήματα, για ποιον ακριβή στόχο. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι λεπτομέρειες κύριε Επίτροπε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πραγματική αξιολόγηση εφόσον μάλιστα τα προγράμματα έρευνας 13.000 ερευνητές δηλώνουν ότι έχουν προβλήματα. 13.000 ερευνητέ δηλώνουν ότι θα παρετηθούν από αυτά τα προγράμματα αφού δεν έχουν τις λεπτομέρειες που πρέπει. Και τρίτον, μου φαίνεται ότι η στρατηγική του 2020 είναι πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί όταν δεν αφού δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι γενικές συνθήκες που θα ισχύουν μέχρι τότε. Αυξάνεται ο ρόλος της Ασίας, αλλάζουν οι αγορές γενικότερα δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο είδους εξωτερικό έγγραφο που να κάνει μια αξιολόγηση του τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη μέχρι το 2020, εξωτερικές προοπτικές. Αυτό δεν θα άλλαζε υποχρεωτικά ολόκληρη τη δομή της μεταρρύθμισής σας, αλλά ίσως να έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε για αυτές τις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η Άννα Γένσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, Επίτροπο που ήρθε ε, εδώ. Είναι ενδιαφέρον ε, το έγγραφο και ακόμη περισσότερο το παράρτημα και υπάρχουν πολύ καλές ιδέες που αναφέρονται. Αλλά αυτό που μας λέτε είναι μία αντιμετώπιση βήμα προς βήμα και μία προσέγγιση ε, για κάθε χρόνο ε, ανανεωνόμενη. Είναι όμως σωστό, ε, δεν έχετε κανένα προγραμματισμό από τώρα μέχρι το 2014, δηλαδή δεν ξέρετε τι θα γίνει με, το, με τους στόχους της Λισαβόνας και πώς θα μπορούσαμε ίσως να μεταφέρουμε πόρους από προγράμματα που δεν λειτουργούν προς προγράμματα που λειτουργούν ε, διότι θα ήθελα επισήμως να μας πείτε τι γίνεται. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου το 2012 και 2013 δεν θα βοηθηθούμε από τους πόρους του τομέα της γεωργίας. Ε, δηλαδή εκεί ε, δεν θα υπάρχουν πόροι που δεν θα δαπανηθούν. Δεν έχουμε αυτή την ευελιξία. Οπότε γιατί δεν μας λέτε ποια είναι η ουσιαστική αναθεώρηση των ε, ισχυουσών ε, δημοσιονομικών προοπτικών καθώς επίσης και μερικές ιδέες για αναθεώρηση ώστε τα δύο-τρία επόμενα χρόνια να μπορούμε να δράσουμε αντί να καθόμαστε με στραβερωμένα χέρια. Είναι, ε, υπάρχει όντως αυτή η έλλειψη φιλοδοξίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν θέλει να κάνει τίποτα δημοσιονομικά όσον αφορά τη δημοσιονομική προοπτική μέχρι ότου φτάσει εντάσσεται στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική και στην επόμενη επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να μπορέσω να συζητήσουμε, ε, θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και από τη σκοπιά της Επιτροπής Δικαιοσύνης. Ε, μιλάμε για την ευρωπαϊκή πολιτική μέχρι το 2020 και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν ε, για το μέλλον και ε, σχετικά με τις συζητήσεις για τους ίδιους πόρους μία συζήτηση η οποία επαναλαμβάνεται σε αυτή την Επιτροπή και επιπλέον ε, μιλάμε για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ιδίως όσον αφορά την διάρκεια του 5 συν 5 που είναι η τελευταία ιδέα στη μόδα και επιπλέον υπάρχουν και τα αρνητικά στοιχεία αυτού του εγγράφου στις ιδέες των 5 συν 5. 5 συν 5 είναι μια εξαιρετική πρόταση αρκεί η αναθεώρηση στα μέσα της διαδρομής να είναι όντως αναθεώρηση η οποία θα εισακούσει τις επιθυμίες μας και θα αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο αυτό. Εγώ δεν ήμουν εδώ όταν διαπραγματευτήκατε τις προηγούμενες προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές αλλά από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι όταν οι προοπτικές αυτές είχαν ε, ε, υιοθετηθεί ξέραμε ότι θα υπήρχαν προβλήματα χρηματοδότησης γι' αυτό και συμφωνήσαμε να υπάρχει αναθεώρηση στο μέσο της διαδρομής για να δούμε τι λειτουργήσε καλά, τι λιγότερο καλά, τι δεν λειτουργεί καθόλου και ε, να διαθέσουμε για τα πράγματα που δεν πάνε τόσο καλά περισσότερους πόρους. Οπότε Οπότε ε, θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα λύσουμε δηλαδή τα προβλήματα χρηματοδότησης που έχουμε ήδη, διότι το έγγραφο αυτό μπορεί όντως να χρησιμοποιηθεί για την επόμενη δημοσιονομική πολιτική, χωρίς όμως να λύνει τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Συμμετέχουμε στους κανόν, εσείς συμμετέχετε ή στις συνδιαλλαγές και ή στους τριμερείς διαλόγους, ξέρετε ποιες είναι οι ανησυχίες μας και αυτό που με ανησυχεί επιπλέον είναι η έλλειψη φιλοδοξίας, ότι ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε το έγγραφο αυτό δύο χρόνια αργότερα, δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να ξέρουμε τώρα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο το έγγραφο αυτό, το οποίο είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι και το καλύτερο, έχει κάτι άλλο να μας προτείνει. Ο κύριος Λάσλος Σούριαν. Ευχαριστώ. Ε, έχω να κάνω δύο σχόλια. Η ο Επίτροπος μας είπε ότι η Επιτροπή είχε δύο στόχους όσον αφορά την πολιτική ε, συνοχής. Καταρχήν να λύσουμε τα προβλήματα των γεωργών που είχαν προβλήματα. Ξαναξεκινώ για τρίτη φορά. Ο ένας στόχος ε, της πολιτικής συνοχής ήταν να βοηθήσουμε τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ε, αναπτύξουμε παραδείγματος χάρη ε, της πόλης θα ήθελα να τονίσω ότι η πολιτική συνοχής ε, είναι μία από τις επιτυχημένες ιστορίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει όμως να πούμε ότι παρόλα αυτά υπάρχει μία ανεφροηγουμένου διαφορά μεταξύ των πολύ ανεπτυγμένων περιοχών και των περιοχών που καθυστερούν να αναπτυχθούν. Εάν λοιπόν αλλάξουμε αυτή την πολιτική θα εγκαταλείψουμε την αρχική μας πρόθεση και θα είμαστε ενάντια ε, την αλληλεγγύη που πρέπει να διέπει εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μία σύντομη μνήα εις τα προβλήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον στο έγγραφο αυτό και ότι πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε την ε, ρήπανση αλλά αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν ε, στο ποδάρι ή εις βάρος των προγραμμάτων που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ακούσαμε τον κύριο Μπαρόζο που μιλούσε για μία λύση υπό τη μορφή 5 συν 5 και ορισμένοι ε, τρόμαξαν με ε, αυτήν την ε, προπτική οι άλλοι, οι άλλοι όμως τη θεωρούν ορθολογιστική και πιστεύουν ότι ενδεχομένως είναι και λογική αρκεί στα μέσα της διαδρομής να γίνει μία πραγματική αναθεώρηση και όχι μία υποτυπώδης όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Πίτροπε πόσο εσείς διαβλέπετε την μετάβαση από ένα σύστημα επτά ετές σε ένα σύστημα το οποίο ε, θα βασίζεται στη λογική των 5 συν 5 ετών διότι δεν μπορούμε μετά από 14 χρόνια να εφαρμόσουμε 10 χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Τι διαβλέπετε σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ κύριο Πόρτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, έχω μιλήσει στην Επιτροπή ήδη για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών και μένω στις θέσεις που εξέφρασα τότε. Θα ήθελα να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Το έγγραφο αυτό ενέχει κάποιες ενδιαφέρουσες ε, ιδέες. Θα μπορούσαν να ε, το αποκαλέσω ένα έγγραφο που μας οδηγεί προς τα ε, μπροστά. Τι εννοώ εργαζόμαστε για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Πολύ περισσότερο από το να κάνουμε μία συζήτηση για ιδέες σχετικά με την αναθεώρηση των ε, ισχύουσων ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Λοιπόν, μιλάμε για τις μελλοντικές προοπτικές, ενώ ε, βιώνουμε μία περίοδο αυστηρής λιτότητας. Εάν ταυτόχρονα δεν καταφέρουμε να συζητήσουμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση των τωρινών προοπτικών, τι σημαίνει αυτό. Μολύνουμε, ρηπαίνουμε το μέλλον με βραχυπρόθεσμες, κοντόφελμες πολιτικές επιλογές. Αυτό ε, ε, είναι και η αδυναμία αυτού του εγγράφου κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή τι, κάνουμε ένα άλμα και πηδάμε στο μέλλον ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του 2012 και 2013. Αυτή είναι η επίπτωση. Δηλαδή, εάν δεν πάρουμε στα σοβαρά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα το 2012 και 2013, είναι προφανές ότι ε, το 2014 εμείς ε, θα παρατείνουμε την κρίση για το επόμενο πολιετές πλαίσιο. Δεύτερη παρατήρηση. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν πως χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό σαν αντιστάθμιση των προβλημάτων του νομίσματος. Συγγνώμη, αυτό τη δεκαετία του 80 όταν δημιουργήσουμε τη, τις πολιτικές συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία ήταν σαφές. Αλλά είναι σίγουρο ότι ε, με, το οικονομικό κλίμα, το οικονομικό πλαίσιο, όχι η συγκυρία, έτσι, το οικονομικό πλαίσιο που επικρατεί, ε, σαφώς διαφέρει από αυτό της δεκαετίας του 80. Μία πτυχή του είναι η εξή. Ότι έχουν αποκλίνει οι ρότε των χωρών. Έχουμε τι χώρε τι πλεονασματικέ και τι ελληνικέ. Και ανάμεσά του άνοιξε ένα χάσμα, ένα γκρεμό που συνεχώ διευρύνεται. Και εξάλλου αυτό ε, αντανακλά και το χάσμα των κοινωνιών μας, ε, αντανακλά την κοινωνική ανισότητα. Τη δεκαετία του 90, χάρη στις πολιτικές ε, συνοχής, και αυτό ήταν ο στόχος τους κιόλας, μπόρεσαν οι περιφερειακές χώρες, οι ουραγοί της Ένωσης να αναπτυχθούν ταχύτερα σε σχέση με τις χώρες του κέντρου. Αυτή η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θέτει μία τελεία ε, ε, ε, και παύλα στις δυνατότητες αυτού του προτύπου. Πλέον δεν είναι σε θέση αυτό το πρότυπο να καλύψει ούτε αυτό το χάσμα ούτε και να ε, καταπολεμήσει τις επιπτώσεις των κοινωνικών δυσκολιών. Γιατί και αυτό ήταν ένας από τους στόχους ε, της πολιτικής συνοχής. Ε, δηλαδή αυτά τα προβλήματα που συνιστούν το πυρήνα της σημερινής περίοδου δεν αντιμετωπίζονται από αυτό το έγγραφο. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν, δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται και έχω αμφιβολίες. τα τελευταία χρόνια είχα τη δυνατότητα να συζητήσω τα θέματα αυτά με τον Επίτροπο Λεβαντόσκι και πολλές φορές μου είπε ότι είμαι πολύ ανυπόμονη διότι το 2006 όταν συζητήσαμε τις τωρινές δημοσιονομικές προοπτικές είχαμε διαπραγματευτεί μία ότι θα υπάρξει μια ισορροπημένη εξέλιξη διότι πιστεύαμε ότι γρήγορα πρέπει να αλλάξει κάτι ώστε να είμαστε πιο επιτυχείς οικονομικά και πολιτικά. Ορισμένοι ε, πήγαν την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα όπου είναι τώρα ε, η αγορά για την αιωλική ενέργεια. Ε, προχωρούν επίσης πάρα πολύ με την ηλιακή ενέργεια. Οπότε δεν πρέπει να τους αφήσουμε την κυριαρχία σε τέτοια συστήματα. Αυτό έχει σημασία και με την ε, στρατηγική μας ε, προοπτική για τη βιομηχανική πολιτική. Σκέφτομαι λοιπόν την ε, προοπτική του 2020 και αναρωτιέμαι πώς αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό και ιδίως και για το 12 και για το 13 και ιδίως για το 14. Οπότε το έγγραφο αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο πολύ ένα έγγραφο συλλογιστικής και όχι ουσιαστικά παρεμβάσεως από ότι, αντιθέτως σε ό,τι είχαμε συμφωνήσει και επίσης στο Συμβούλιο αντιλαμβάνομαι ότι τα κράτη-μέλη ε, ε, πάντοτε λειτουργούν πιο διακυβερνητικά το οποίο δεν πρέπει να είναι καλό ούτε για μας ούτε για σας. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι τι πολιτική συνέπεια εσείς ε, μπορείτε να αποκομίσετε και τι σκοπεύετε να κάνετε για να προασπίσετε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ κύριος Μπέγκερ. Ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω με όσα είπε η Έλγα ε, διότι υπάρχει κίνδυνος ε, να ε, οπισθοδρομήσουμε στην κατάσταση πρώτης Λισαβόνος πράγμα το οποίο είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Είχαμε όντως ορισμένες υποσχέσεις από το έγγραφο της Επιτροπής. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο αναμέναμε. Ε, περιμέναμε πολύ περισσότερα και στο έγγραφο αυτό υπάρχουν μεν ορισμένες ενδιαφέρουσες ε, ε, συζητήσεις τις οποίες είχαμε και τότε και που ε, επιτρέπουν επιπλέον να προχωρήσουμε στις δημοσιονομικές προοπτικές. Αλλά όπως είπε η Έλγκα, όλα αυτά είναι ωραία ως ασκήσεις επί χάρτου, αλλά τι θα γίνει περί του πρακτέου. Και έχω δύο ερωτήσεις προς τον Επίτροπο. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, στο έγγραφο η Επιτροπή αναφέρεται σαφώς σε μία σειρά ενδιαφερουσών δυνατοτήτων για να προχωρήσουμε και λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον κατάλογο που δεν είναι πλήρης <clears throat> θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να προτείνει ε, ίδιους πόρους οι οποίοι θα επιτρέψουν μία βαθμιαία μείωση των ε, συνδρομών των κρατών μελών. Αλλά ε, δεν θεωρώ ότι ο κατάλογος αυτός είναι πλήρης και μπορεί να προχωρήσει Χρειάζονται ακόμη προσθήκες και κάποια δεδομένη στιγμή θα πρέπει να δούμε τι είναι οι δυνατότητες και τι σημαίνουν για τους ίδιους πόρους. Δηλαδή, ε, μία πρόταση. Πρέπει να αναλάβετε την ε, πρωτοβουλία. Έχετε το δικαίωμα πρωτοβουλίας και πρέπει να υποφεληθείτε. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το δικαίωμα της πρωτοβουλίας εάν δεν το χρησιμοποιούμε. Είναι το ίδιο με το Συμβούλιο όπου υπάρχουν ε, τα ειδικά συμβούλια και θέματα που έπρεπε να ε, λύσουν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνονται από το Συμβούλιο και τότε βέβαια διαπιστώνουμε ότι όντως η Επιτροπή δεν έχει την πρωτοβουλία και έχει τώρα την ευκαιρία να κάνει κάτι σχετικά με αυτά που βλέπουμε στο έγγραφο αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχουμε ουσιαστικά τρία πρότυπα και τρία μοντέλα στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν, ε, ε, βάσει μίας εκθέσεως κατά πρωτοβουλία είχε γίνει μία συζήτηση για μία ε, δυνητική επέκταση σχετικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας για να ακολουθήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα είναι δημοκρατικά πιο ε, νομιμοποιημένο. Υπάρχουν επίσης συζητήσεις όπου λέγεται ότι θα φτάσουμε στα πέντε χρόνια καταρχήν ε, παρατείνοντας ως τα πέντε χρόνια και ίσως ε, πρέπει να καταπιούμε για μια ακόμη φορά από πλευράς του Συμβουλίου την επταετία και μετά θα πάμε στα πέντε χρόνια και μετά θα έχουμε τα πέντε συν πέντε και διαμέσως θα υπάρχει υπάρχει ένα κενό. Αν μιλάμε λοιπόν για ένα τέτοιο πρότυπο όπου βλέπω τα κράτη μέλες, ιδίως ε, τα κράτη ε, ε μέλη ε, θα μπορέσουν ε, να υποφεληθούν ε, πόρων που έχουν προβλεφθεί για μία δεκαετία τότε ακόμη και η δικιά μου περιφέρεια θα συμφωνήσει αλλά τότε θα δούμε ότι δεν ελέγχουμε κάθε 5 ή 7 χρόνια αλλά κάθε 10 χρόνια και οι συνολικές απαιτήσει για έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις ε, θα κατέρε. Και γι' αυτό Πιστεύω κύριε Επίτροπε και εδώ σκέφτομαι την Γιούτα και το Σαλβαντόρο ε, και θέλω να σκεφτούμε ε, τι είναι οι κίνδυνοι αυτών των προτύπων. Πιστεύω ότι όσο πιο δυσμενείς είναι η αριθμή τόσο λιγότερη πρέπει να είναι η διάρκεια και όσο πιο ε, ανικανοποιητικά ε, είναι η δυνατότητα ευελιξίας τόσο λιγότερο πρέπει να είναι και ο χρόνος διαρκειάς τους. Οπότε ε, όταν μιλάμε για την επιστολή των 6 ε, την οποία ζητούμε να υιοθετήσουμε νομίζω ότι αυτή είχε υποβληθεί το Δεκέμβριο του 2004 ή κάτι τέτοιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, ήδη τα 5 συν 5 δηλαδή με την αναθεώρηση είναι ήδη πεπερασμένα και το Κοινοβούλιο δεν θα το δεχθεί αυτό ποτέ. Διαφορετικά εμείς μόνοι μας θα βγάλουμε τα ίδια μας τα μάτια και θα αποκλειστούμε από την ε, ε, πολιτική διαπραγμάτευση. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε αυτά τα οποία όντως ε, είναι υλοποιήσιμα σε πολιτικό επίπεδο και μετά να αποφασίσουμε για την διάρκεια συγκεκριμένων ενεργειών. Δηλαδή, αν έχουμε τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον ε, μία μειοψηφία που μπλοκάρει ότι καλύτερα είναι να παραμείνουμε ε, σε αυτά τα οποία ε, θα θέλαμε, τότε καλό θα ήταν όντως να παραμείνουμε εκεί που βρισκόμαστε τώρα. Εάν υπάρξουν λοιπόν προσαρμογές και βελτιώσεις για την Λισαβόνα, δεν μπορούμε τώρα να προεξοφλήσουμε πώς θα ε, τις αντιμετωπίσουν ορισμένα κράτη-μέλη διότι ε, παραδείγματος ε, χάριν, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πακέτο σταθερότητος εκτός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και έτσι θα πούμε ότι με κάτι τέτοια μέτρα και με στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας προχωράμε, τουλάχιστον δίνουμε μία καλή εικόνα στο δημόσιο, αλλά τότε έχουμε εγκαταλείψει την προοπτική 5 συν 5 και γι' αυτό όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αρνείται ε, μία πρόταση κατά πρωτοβουλία, δεν νομίζω ότι πράττει σωστά. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να έχουμε ε, υπολογίσει ποια είναι τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων προτύπων που προωθούνται, να παρακολουθούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και η συζήτηση αυτή ε, να ε, επανέλθει ε, στις αρχές του χρόνου στην Επιτροπή την Αρμόδια ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Έχουν ακόμη πολύ ζητήσει το λόγο. Ένα λεπτό στον καθένα. Γιατί αλλιώς δεν θα προλάβει να απαντήσει ο Επίτροπος. Λοιπόν, ο Αντιπρόεδρος Αλβάρος. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι θα μου αρκέσει ένα λεπτό. Θέλω να απαντήσω σε αυτά που είπε η συνάδελφος Αν Γένσεν. Η αναθεώρηση που αναμένουμε, τι στοχεύει. Το μέλλον, αλλά βέβαια θα βασίζεται και στο παρελθόν ως εμπειρία. Θα ήθελα λοιπόν κάποια πληροφόρηση επ' αυτού πώς γίνεται ακριβώς η δαπάνηση του προϋπολογισμού. Γιατί αν απλώς ζητούμε όλο και περισσότερα χρήματα πρέπει να ξέρουμε και πώς ακριβώς δαπανώνται. Δεν έχω δει καμία μελέτη που να λέει ποια είναι η προστιθέμενη αξία ενός ενωσιακού ευρώ. Αφού προγραμματίζουμε το μέλλον πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματικά δαπανίσαμε τα χρήματά μας στο παρελθόν. Ευχαριστώ αγαπητέ μου συνάδελφε, η κυρία Αντιπρόεδρος Ούτελχάου της Επιτροπής ΣΟΥΡ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πρόκειται για προοπτικές που θα πάνε πολύ μακριά στο μέλλον αναγκαστικά. Πέντε χρόνια ας πούμε. 14 με 18. Γιατί είναι πολύ πιθανό Εξάλλου, οποιαδήποτε περίοδο και να θέσουμε, μακρά ή όχι, να μας λείψουν τα χρήματα τελικά. Αλλά υπάρχει η κοινοτική ενωσιακή βάση που τη δέχτηκαν και η Κομισιόν και το Συμβούλιο με βάση μια πολύ θετική αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο, δηλαδή τη στρατηγική του 2020. Η στρατηγική αυτή πρέπει να τη δούμε τη στρατηγική αυτή σφαιρικά το είπαμε και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε. Δεν πρέπει να ζητάμε από όλες τις γενικές διευθύνσεις αναγκαστικά να συμφωνήσουν πρώτα μεταξύ τους, αλλά μάλλον να συνδέσουμε το εθνικό επίπεδο με το ενωσιακό τιούτο. Και για να γίνει κάτι τέτοιο υπάρχει μια σταθερή και γνωστή βάση. την οποία έχουμε πει πολλές φορές στο έγγραφό μας, εδώ, τι προτείνουν. Προτείνουν μια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και τα λοιπά. Και τα λοιπά Αν θέλουμε ιδιαίτερα να αναφερθούμε στο λειτουργικό πρόγραμμα σε περιφερειακό επίπεδο όπως προτείνει η Κομισιόν και επί του οποίου ζητάει βελτιώσεις, αν βασιστούμε σε αυτό λοιπόν, μάλλον αν το αγνοήσουμε αυτό, περί τίνος άλλου πρόκειται. Πρέπει να δούμε τι δυνατότητες έχουμε για πληροφόρηση και θα δούμε τι γίνεται με το κρέας και αν θα είναι ευρωπαϊκό κρέας παρόλο που πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι η υπεύθυνη για τη γενική πολιτική και για το σκελετό ε, δηλαδή για το τι πρόκειται να, ε, να, βασί, να ε, προωθήσει το σκελετό υπεύθυνα είναι τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Γκέραν Χέρμ. Ευχαριστώ. Κάποιες σκέψεις μόνο, Πρόεδρε. Αν κάποια κράτη-μέλη είναι σοβαρά όταν κάνουν την εξή πρόταση, δηλαδή να μειώσουν στο 0,8% τον επόμενο προπολογισμό, στο επόμενο πλαίσιο. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, θα χάσουμε γύρω στα 30 δίσε από το δικό μας τον προπολογισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα βασικά στοιχεία. Τι θα γίνει αν κόψουμε, περικόψουμε 30 δις από τον ε, προϋπολογισμό της Ένωσης. Μιλάμε για προστιθέμενη αξία της ε, Ευρώπης, ε, αλλά συγγνώμη φαίνονται κρίσιμα τα ζητήματα. Δεν... Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Ο James Ellis είπε ότι 30.000 ερευνητές καταγγέλουν την γραφειοκρατία στο ερευνητικό πλαίσιο. Ακόμη χειρότερο είναι ότι έχουμε 300-400.000 ερευνητές στην Ευρώπη, εκτός Ευρώπης, διότι δεν μπορούν να βρουν ένα καλό μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τον προπολογισμό τη Ένωση και να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου προβλήματα. Α θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να αποδείξουμε γιατί είμαστε ικανοί για την εσωτερική αγορά, παραδείγματο χάρη. Γιατί αποτύχαμε και δεν οικοδομήσαμε μια πραγματική ε, εσωτερική αγορά. Δεν μπορέσαμε, παραδείγματο χάρη, να έχουμε σιδηροδρομική υποδομή, ενεργειακή υποδομή που να συνδέει όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Αν είμαστε σε θέση να το κάνουμε, τι θα συνεπαγόταν αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα βασικά ζητήματα εδώ κατά τη γνώμη μου και να ε, περιγράψουμε τη διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και στη μη Ευρώπη. Ε, γιατί στη μη Ευρώπη θα καταλήξουμε αν κόψουμε 30 δις από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Επίσης πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ε, έχουμε χρήστη, να, μάλλον να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά ε, τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Εντάξει, ωραίο αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία. Πολύ ωραία ιδέα, αλλά πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Το ελεγκτικό συνέδριο ακόμη κατακρίνει ε, τι επιδόσει των διαρθρωτικών ταμείων. Υπάρχουν πολλά πράγματα, τα είπατε κι εσείς, ε, ε, ε, ξεκινούν αργά τα προγράμματα, είναι περίπλοκα τα πράγματα, υπάρχει γραφειοκρατία. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με σήμερα, αλλιώς δεν θα απορροφηθούν τα κονδύλια από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να ε, ασχοληθούμε με τα βασικότερα ζητήματα. Αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Ε, Γεωράν, ο κύριο Γκότμανης, σύντομα. Κοιτάζω το λεπτό για να σεβαστώ το ένα λεπτό. Ε, τρία λεπτά θέλω να πω. Αν αναλύσει, Αν κανείς τον προϋπολογισμό του 11, βλέπει ποιοι κίνδυνοι εμπεριέχονται. Πρώτον, από πού προέρχονται τα χρήματα για το διορθωτικό προϋπολογισμό οι αναπτυξιακοί κανόνες δεν είναι σαφείς. 1,7 δισεκατομμύρια το πέρυσι δεν δαπανήθηκαν. Πρέπει να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πρόκειται εδώ για μια πηγή χρημάτων που δεν χρησιμοποιείται. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεύτερον, η πολιτική συνοχή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 5 και 5 ή για 10 χρόνια κτλ. Διότι αν δούμε τις ε, ανηλυμένες μας υποχρεώσεις, τις προβλεπόμενες δαπάνες, βλέπουμε ότι δεν καταλήγουν σε πληρωμές παρά με μεγάλη καθυστέρηση. Τον πρώτο, το δεύτερο, τον τρίτο χρόνο μόνο κατέληξαν σε πληρωμές. Θα βλέπει κανείς λοιπόν εύκολα ότι χρησιμοποιούνται τα χρήματα για άλλους στόχους από όσους έχουν προβλεφθεί. Και μας είπατε κύριε Επίτροπε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα της μη απορροφητικότητας. Και αφού υπάρχει κάτι δεν πάει καλά. Χορηγούνται χρήματα και σε πληρωμές χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πώς κυμαίνεται η πραγματική χρήση συν 13, συν 15, 5 και 5. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα γιατί στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση τι βλέπουμε ότι στον πέμπτο χρόνο μόνο 70% έχει απορροφηθεί. Για να φτάσουμε στο 100% δεν χρειάζονται 7 χρόνια αλλά κάτι σαν 11. Άρα τελικά δεν θα μπορέσουμε να το δούμε συνολικά όπως θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος, ο κύριος Ιβο Κάλφη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα, uh, what you... έχει ζητηθεί επανειλημμένως μεγαλύτερη συνοχή στον προϋπολογισμό. και καλύτερη χρήση και βελτίωση γενικότερα της απορροφητικότητας. Πώς ακριβώς θα το πετύχουμε αυτό δεν ξέρουμε. Ερωτώ λοιπόν, δεν πρέπει να δούμε και τι θα χάσουμε από αυτά τα μέτρα. Καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να κάνει μια έκθεση για το κόστος της μη Ευρώπης, αλλά δεν μπορεί να κάνει μια έκθεση όχι για την μη Ευρώπη αλλά για την λιγότερη Ευρώπη που είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στον προϋπολογισμό. Εγώ θα έλεγα ότι η συμπερίληψη του κριτηρίου της σταθερότητας στην Ευρωζώνη θα ήταν κάτι που θα κατέληγε σε πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα αλλά δεν μιλάω καν για τις δαπάνες. Ο ρόλος του προϋπολογισμού λοιπόν είναι κάτι που δεν πρέπει να το περιορίσουμε σε έκφραση ωραίων ιδεών, ευρωομολόγων και τέτοια, αλλά πρέπει να δούμε λίγο γενικότερα στο μέλλον τι χάνουμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Σας ε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μία παρατήρηση θα κάνω μόνο εγώ. Αναθεώρηση πίτροπε. μια, λοιπόν, έναν ορίζοντα δεκαετή. Ε, ας έχουμε το θάρρος ε, να παραδεχτούμε το εξής. Η... Λισαβόνα έχει προβλέψει 10 χρόνια για το στόχο της ανταγωνιστικότητας και τι, ήταν 10 χρόνια ονειρικά. Ε, η στρατηγική Ευρώπη 2020 όμως πρέπει να μην είναι ονειρική, πρέπει να είναι πραγματική. Ε, αυτό απαιτεί να βρούμε τα μέσα και για να χρηματοδοτήσουμε τις ε, κοινωτικές πολιτικές μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, άρα χρειάζονται νέα κονδύλια. Επίσης θα πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα συμβάλλουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί για να χρηματοδοτήσουμε τους κοινούς στόχους της Ένωσης. Ε, ορισμένα πράγματα χρηματοδοτούμε μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά πάλι δεν μπορούν να υλοποιηθούν παρά μόνο χάρη στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η δεκαετία που ξεκινάει τώρα θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να χαρακτηριστεί από το εξής. Ε, από την στενή συνεργασία του, των εθνικών προϋπολογισμών με τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτό είναι ένα κεκτημένο για την εξυγίανση των δημοσιονομικών, την καταπολέμηση των χρεών, των ελλημάτων κτλ. Μέσα από την οικονομική διακυβέρνηση. Δηλαδή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Αυτό τώρα που θα χρειαστεί για την ε, υλοποίηση του ε, ε, μηχανισμού χρηματοπιστωτικής στήριξης θα είναι η χρηματοδότηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει χρηματοδότηση για αυτό το μηχανισμό και πρέπει να το ρυθμίσουμε το ζήτημα. Πρέπει να έχουμε δε κατά νου πως η διαδικασία αυτή έχει νόημα μόνο αν είμαστε σε θέση με κάποιον τρόπο που θα τον βρούμε εμείς ε, να ε, ε, αποκτήσουμε μεγαλύτερες συνεισφορές από πλευράς των εθνικών προϋπολογισμών. Ναι, Επίτροπος. Ευχαριστώ. έχουμε, ακούσαμε την παρουσίαση, έγινε συζήτηση. Ε, με όλες αυτές τις ερωτήσεις που άκουσα είναι απαιτητική η συζήτηση και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διαθέσή μας. Ε, εν είδη γενικής παρατήρησης θα έλεγα ότι κατά τη γνώμη σας δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και δεν πρόκειται για να αναθεώρηση των τωρινών δημοσιονομικών προοπτικών, είναι ένα μόνο έγγραφο προβληματισμού. Ναι, είναι και έγγραφο προβληματισμού. Δεν ποσοτικοποιούμε ε, τις επιπρόσθετες ανάγκες που θα έχουμε ε, για την περίοδο 2011 ως 2013 ε, υπάρχει κάποια ποσοτικοποίηση σε σχέση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 όπως είπατε, αλλά αυτό είναι λίγο παραπάνω από το 40% του τωρινού προϋπολογισμού και πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τη στρατηγική 2020. Ε, είναι θεμητή η επίκριση που μας απευθύνεται. Δεν πρόκειται για αναθεώρηση των τωρινών προοπτικών και όπως είπαν σχεδόν όλα τα μέλη της κόμπου Πρόκειται για πολιτική δήλωση, ο Ράιμαρ Μπέγκε και η Χέλμα, Χέλγα Τρουιπέλε έκαναν αυτή την παρατήρωση, οπότε θα δώσω και εγώ πολιτική απάντηση. Ε, υπάρχει ε, κάποια ποσοτικοποίηση των αναγκών μας σήμερα. Ε, και θα ακολουθήσουμε την σταδιακή προσέγγιση για την ποσοτικοποίηση, διότι η βάση των δημοσιονομικών αρχών ε, χρειαζόμαστε μια νομική βάση για να κατανείμουμε τα κονδύλια. Έχουμε την ημερησία εξωτερικής ε, δράσης, σαφώς υπεδείχθη και αυτό είναι στην δήλωση για την ετήσια διαδικασία ότι οι δαπάνες για την κοινή εξωτερική πολιτική διπλασιάζονται σε σχέση με το 2007, το ίδιο για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές ε, υποθέσεις. Χρειάζονται λοιπόν προσαρμογές ε, για να συμφωνήσουμε για το μελλοντικ... μελλοντική αιτήσια διαδικασία, για το ίτερ ή για ε, το μηχανισμό για τις μπανάνες. Χρειαζόμαστε και νομική βάση, εντάξει, ναι κάτι τετριμένο, δεν χρειάζεται ε, να μας απασχολεί αυτό ε, κατά προτεραιότητα. Τι γίνεται τώρα με τη στρατηγική δεδομένων των συμφραζομένων της τωρινής κατάστασης. Έχω την εντύπωση πως ε, έχουμε εισέλθει σε διακυβερνητικά πεδία, Δηλαδή, οι επιπτώσεις ε, της Λισαβόνας ε, δεν επηρεάζουν αυτούς που σχεδίασαν ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας μόνο, αλλά συνδέονται άμεσα με την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη. Ο στόχος μας ήταν να μην προκαλέσουμε υπερβολικά, να εισηγηθούμε μια, έναν ισόρροπο προϋπολογισμό, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ασχολούμενοι με τα έσοδα Έχουμε το οικονομικό μείγμα ε, της αποταμίευσης με αυξημένη φορολογία. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη και ήδη προκαλούμε αρκετά με αυτά. Δηλαδή το σύνηθες οικονομικό μείγμα που ακολουθείται σε περίπτωση εξυγίανσης των δημοσιοοικονομικών, αυτό υπαγορεύει, δηλαδή επιπρόσθετους φόρους και όχι αυξημένες εισφορές στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ήδη προκαλούμε ε, αυτό και σας μιλώ για το σύστημα των ιδίων πόρων, Ε, τώρα θα κάνω μία πολιτική παρατήρηση για τη στρατηγική του Κοινοβουλίου. Δεν θέλουμε τον ε, Δεκέμβρη να προκαλέσουμε υπερβολικά στη Σύνοδο, δηλαδή στις Βρυξέλλες. Θέλουμε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα της Επιτροπής ε, να υποβάλει με αυτόνομο τρόπο ρεαλιστικές και φιλόδοξες προτάσεις για την περίοδο μετά το 2013. Εάν το σκοτώσουμε εθνισυγενές το σχέδιο, ε, αν ε, το σκοτώσουμε εξ αρχής στο σχέδιο, ε, θα θεωρείται ότι μαγειρεύουμε εκ των προτέρων. In being realistic. και ξαναλέω πρέπει να είμαστε ρεαλιστές από πολιτικής πλευράς όταν παρουσιάζουμε το όραμά μας για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Είναι συνειδητή η επιλογή μας ε, δηλαδή. Σας απογοητεύουμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και το Συμβούλιο. Ας ελπίσουμε ότι η διαδικασία σύνδεση του ετησίου προϋπολογισμού με την αναθεώρησή του από κοινοβουλευτικής πλευράς ε, δεν θα προδικάσει την έκβαση της Συνόδου του Δεκεμβρίου. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά ας το ελπίσουμε γιατί εδώ μιλάμε για την πολιτική εμπλοκή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία και προφανώς είναι ευπρόσδεκτη η παρουσία του Κοινοβουλίου στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα είναι ένα αξιόλογο επίτευγμα, αν καταστεί εφικτό. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφής δήλωση το Δεκέμβριο. Φοβούμε μήπως περιοριστούμε τελικά εάν δεν έχουμε μία ρεαλιστική προσέγγιση για τον προϋπολογισμό μετά το 2013. Αυτή είναι η πολιτική αιτιολόγηση της ε, συνετής προσέγγισης μας, ε, δηλαδή να παρουσιάσουμε την αναθεώρηση χωρίς να έχουμε πλήρη ποσοτικοποίηση των επιπροσθέτων αναγκών, ε, κυρίως όταν μιλάμε για νέα κονδύλια διότι μέσω της ανακατανομής έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το Ήτρε, για τις μπανάνες, για τις υπόλοιπες δαπάνες, για την Παλαιστίνη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανακατανομή των κονδυλίων, να ε, ζητήσουμε το μέσο ευελιξίας μόνο όταν χρειάζεται. Αυτή είναι η πιο βασική επιφύλαξη που έχετε, το βασικό συνδυασμό που έχετε και άρα δίνω πολιτική απάντηση σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν. Και αν διαβάσετε και το τεχνικό παράρτημα θα δείτε στο μέλλον ε, πώς έχουν ε, οι δαπάνες ε, σε διάφορους τομείς πέρα από τους ίδιους σπόρους. Έτσι όλα τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πακέτο που θα υποβληθεί του χρόνου. Αυτά για την ε, ε, ε, κατηγορία που μας απαγγείλατε και θα σας απαντούσα ότι πρέπει να είμαστε και πολιτικοί και όχι μόνο τεχνικοί όταν συζητούμε αυτά τα θέματα. Ας περάσω τώρα σε κάποια σε κάποιες πιο τεχνικές παρατηρήσεις. Ο Σαλβαντόρ Γκαρίγκα ζητά σαφώς κάτι παραπάνω από ένα έγγραφο προβληματισμού και με ρώτησε ε, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η πραγματική απλούστευση. Αυτό δεν είναι το αντικείμενο του εγγράφου αυτού. Έχουμε την αθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και ο James Ellis σχολίασε το ίδιο ζήτημα που παραπονέθηκε ότι οι ερευνητές ε, δεν ε, είναι έτοιμοι για να δεχτούν αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία και μίλησε για τους ερευνητές, για τους επιστήμονες και για τους επιχειρηματίες σε δύο κατηγορίες δικαιούχων που υποβάλλουν και τα περισσότερα παράπονα. Και κυρίως όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφενός και αφετέρου ε, οι επιστήμονες και οι ερευνητές. είναι, αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες δικαιούχων και είναι σαφείς οι προτάσεις, αλλά τοποθετούνται στην ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού και θα έλεγα ότι πρέπει να ε, εστιάζουμε την προσοχή μας στα αποτελέσματα, όχι στην εισφορά. Δηλαδή να μην ασχολούμαστε μόνο με τον έλεγχο, μην ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση ε, όταν μιλάμε για το μέσο κόστος, για τα κατακοποκοπή ποσά, ε, για τις για το συντελεστή επιστροφής εξόδων. Όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία θα ανήκουν στη διαπραγμάτευση που θα γίνει μελλοντικά. Πρέπει να δεχτούν πιο γραφειοκρατικές διαδικασίες οι δικαιούχοι. Αυτό αφενός αφετέρου έχουμε και το θέμα της εθνικής διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων. Δίκιο έχετε Υπάρχουν ακόμη παράπονα από το ελεγκτικό ε, συνέδριο, ίσως φέτος να σημειωθεί μείωση με την ε, πολιτική συνοχής. Χρειαζόμαστε ίσως εθνική ε, εξασφάλιση, εθνική δήλωση, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει με τι γεωργικέ δαπάνε, κυρίω σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Πάντω, για την απλούστευση, σα παραπέμπω στην ε, τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, δηλαδή με ποιο τρόπο θα δαπανούμε. Ε, ε, μάθουμε πόσα θα δαπανίσουμε. Γιατί μιλάμε για μια αναθεώρηση που θα καλύψει την περίοδο μετά το 2014. Τώρα, ο Ετζέμι ζήτησε και κάτι άλλο. Μας ρώτησε για τον αντίκτυπο. Μα με αυτά που γνωρίζετε για τον προϋπολογισμό μπορείτε να το δείτε και στην συνολική μεταφορά. Εκεί να βρείτε την απάντηση. Στον διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2010, στη συνολική μεταφορά ε, κονδυλίων. Δεν υλοποιείται πάντοτε, όπως για την ανάπτυξη της υπαίθρου, Υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων που δεν είναι αποτελεσματικά και διαρκώς κάνουμε μεταφορές πιστώσεων προς καλύτερα προγράμματα. Οπότε άτυπα γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου του τρέχοντος προϋπολογισμού. Ε, εν γέννη θα έλεγα ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2010, το πιο σημαντικό του στοιχείο είναι η μείωση κατά ένα δις ε, πάνω κάτω ε, των ε, πληρωμών κάτω από το 1% του προϋπολογισμού. Το 2008 σας είπα ότι είχαμε μείωση κατά 5 δις. Βελτιωνόμαστε δηλαδή ως προς την υλοποίηση του προϋπολογισμού και αυτό είναι και η απάντηση σε αυτούς που θέλουν να τροποποιήσουν τον προϋπολογισμό για τα να απομείνονται έτη ε, των ε, τωρινών δημοσιονομικών προοπτικών. Μα τρέχουν τα προγράμματα και έχουν σχεδιαστεί για ε, κάποια χρόνια και βελτιωνόμαστε και θα δείτε μεγαλύτερη βελτίωση το 2012 και 2013 γιατί δεν έχουμε και με απεριόριστο περιθώριο λιγμών για ανακατανομή των κονδυλίων. Τώρα είμαστε, τρέχουν τα προγράμματα και Είμαστε σε μια κανονική πορεία, κινούμαστε με κανονική ταχύτητα. Ε, ε κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που είπε ο James Ellis. Τι μπορούμε να επιτύχουμε για την ανταγωνιστική, πιο καινοτόμα Ευρώπη. Ωραία. Ε, να αποφύγουμε την διαρροή των εγκεφάλων, όπως λέγει το brain drain. Ε, ο κύριος Άλβαρο το είπε σαφέστατα αυτό και ο κύριος Φάρμα ότι τα, οι καλύτεροι εγκέφαλοι, τα καλύτερα μυαλά φεύγουν από την Ευρώπη. Μα υπάρχουν και όρια στη δράση μας, δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε τις δημόσιες δαπάνες. Ε, παίρνω μια ρητορική στάση, το ξέρω, αλλά αμφιβάλλω προς τους στόχους που θα επιτύχουμε επεκτείνοντας ε, τις δημόσιες δαπάνες ή συγκροτώντας νέα θεσμικά όργανα ή νέους οργανισμούς. Το καινοτόμο πνεύμα έχει σχέση με την κουλτούρα, ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου, το ίδιο με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, αυτά που γίνονται στις χώρες μας. Δεν μπορούμε παρά εν μέρη να αντικαταστήσουμε αυτή την ανάληψη κινδύνου με δημόσιες ε, δαπάνες. Ε, τώρα αυτή είναι η προσωπική μου ε, μάλλον ε, θέση, μια δωρική στάση και βλέπω και τα όρια των φιλοδοξιών μας, ε, των στόχων με, που ενδεχομένως θα επιτευχθούν με επιπρόσθετα κονδύλια συγκροτώντας νέους οργανισμούς για να λύσουμε το πρόβλημα. Μα δεν είναι τρόπος για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της μη καινοτόμας Ευρώπης. Δεν είναι επαρκή απάντηση. Παρόλα αυτά μπορούμε να δώσουμε στήριξη και το είπε και η Έλγα για την καινοτομία και για την ε, κατασκευή νέων πρασίνων τεχνολογιών ε, να χρησιμοποιήσουμε δημόσια κονδύλια. Αυτό γίνεται βέβαια και έγινε και σε πολλές χώρες, σε πολλές υπήρους, αλλά υπάρχουν όρια ξαναλέω ε, σε σχέση με αυτά που μπορείτε μέσω δημοσίων δαπανών να επιτύχετε για την καινοτομία συγκεκριμένα και για την ανταγωνιστικότητα. απάντησα στη γενική κατηγορία ότι τελικά δεν πρόκειται για ουσιαστική ε, αναθεώρηση του προπολογισμού και είναι ένα έγγραφο προβληματισμού. Οπότε τώρα θα ε, σας μιλήσω για τη συνοχή, γιατί ο κύριος Σούριαν σαφώς ε, και ο κύριος Γκοντμάνης, ο κύριος Πόρτες, η Χέλγα, όλοι σαφώς το σχολίασαν και η Γιούτα Χάουγκ. Είναι η κατεξοχήν πολιτική της Ένωση, η πολιτική συνοχής. Ε, για την συνέχιση της πολιτικής υπάρχει καλή επιχειρηματολογία, υπάρχουν καλές δομές, ε, καλή δικαιούχη, αλλά έχουμε και κακές επιδόσεις, έχουμε και κακούς δικαιούχους ε, οι οποίοι διευρύνουν το χάσμα και έχουμε βελόριες δαπάνες και έτσι διευρύνεται το χάσμα. αυτή είναι η αντίεπιχειρηματολογία. Ε, συγκρίνεται όμως το έγγραφο από το 2009 με το έγγραφο αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Θα δείτε μια σαφή διαφορά. Τι λέγαμε το 2009 ε, τότε κάναμε μια τυπική ανακατανομή των κονδυλίων στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Ε, λέγαμε ότι θα επικεντρώσουμε τη συνοχή σε κάποιες συγκεκριμένες τομείς, κυρίως στην Ανατολική, ε, σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, ε, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Τώρα, με τη διόρθωση του προϋπολογισμού θέλουμε να καλύψουμε διάφορες ανάγκες πολιτικής συνοχής. Δεν μιλάμε μόνο για ανακατανομή, θέλουμε να ε, υπάρξει... Να, επέκταση της περιοχής που καλύπτουν τα κονδύλια να ξαναδούμε τα είδη δαπανών, να καλύψουμε τα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν ε, συμπεριλαμβάνονται αυτά καθ' αυτά στην διαδικασία αναθεώρησης, αλλά ε, επισέρχονται στον προβληματισμό του υποφαινομένου και του Επιτρόπου Χάν για το μέλλον της πολιτικής ε, να καλύψουμε ίσως και κάποιες περιοχές της Ισπανίας, ούτως ώστε να έχουμε πολυεπίπεδη πολιτική ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Πρέπει να κάνουμε την επιλογή. Αν θέλετε να επικεντρωθούμε στην ανακατανομητική πολιτική για την Ανατολική Ευρώπη, ε, για την οικογένειά μου από το Ρουμπέλης και στην Πολωνία ή εν πάση περιπτώσει, αυτό θα σημαίνει το τέλος της πολιτικής συνοχής. Έχουμε και άλλες επιλογές. Πρέπει να θεωρούμε ως αναπτυξιακή πολιτική την πολιτική συνοχή ε, και να προωθούμε την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρώπης για τις κακές επιδόσεις και ο κύριος Γκουτμάνης το είπε. Ναι, στην ανάπτυξη της υπαίθρου έχουμε υπερβολική αποταμίευση και πολύ βολικό είναι αυτό να, να κατανέμουμε συνέχεια τα κονδύλια για να κλείσουμε το χάσμα που έχει δημιουργηθεί στο ίτερε. Δηλαδή από πλευράς προγραμματισμού του προϋπολογισμού είναι βολικό αυτό για τα ένα εναπομείνοντα μείνονται των τωρινών ε, προοπτικών. Αυτό είναι ένα είδος αξιολόγηση αντικτύπου ε, σχετικά με την πηγή επιπρόσθετης χρηματοδότησης. Γιούτα Χάουγκ, έχει ασχοληθεί με τη συνοχή και μίλησε ε, για το κρέας. Ε, θέλουμε ε, να συμφωνήσουμε για τις εταιρικές σχέσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ε, σύντομα θα το δείτε αυτό. Σήμερα ακόμη συζητάμε το έγγραφο περί συνοχής και τις επόμενες ημέρες, όχι εβδομάδες, θα δούμε το αποτέλεσμα. Τι κρύβεται από πίσω. Το πνεύμα είναι το εξής. Θέλουμε να απαριθμίσουμε διάφορα εργαλεία συνοχής και να τα ενσωματώσουμε σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπίσουμε την εδαφική διάσταση της συνοχής, δηλαδή να έχουμε πληθώρα εργαλείων υπό μια κοινή αιγίδα, μέσα σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, όταν ε, είναι εφικτό αυτό να έχουμε υποκατηγορίες ε, των εργαλείων συνοχής που ορισμένα θα είναι για την κοινή γεωργική πολιτική παραδείγματος χάρη αλλά η εδαφική ε, χωροταξική διάσταση μας ενδιαφέρει. Διάφορα εργαλεία θα εξυπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο και έτσι θα έχουμε πιο απτά ίσως αποτελέσματα από την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Για να είμαι ειλικρινής, ε, μετά τις επισκέψεις που έκανα σε διάφορες περιοχές και χώρες, κατάλαβα το πιο σημαντικό και επ' αυτού να σας πω ότι χρειάζομαι βοήθεια από το, την Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι το θέμα της ε, συγχρηματοδότησης. Πέρα από την κρίση και την αντιμετώπιση της το 2009 έχουμε και τις ε, ε, προκαταβολές που καταβάλαμε, αλλά τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δίλημα της συγχρηματοδότησης, ούτω ώστε να είναι ρεαλιστική η πολιτική συνοχή. Μιλώντας για το τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για τη συνοχή τίθεται και το ίδιο ζήτημα, γιατί από εκεί ε, προέρχεται προβλέψιμότητα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ο κύριος Μπέγκε ε, είναι ρεαλιστής όταν κάνει αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά τι γίνεται με το 5 συν 5. Ε, θα γώσουν τα, οι αποταμιεύσεις και η λιτότητα, αυτά που ισχύουν τώρα δηλαδή. Δέκα χρόνια ναι μεν, αλλά το εφαλτήριο είναι ότι θα αρχίσουμε το 2011 με μια πραγματική λιτότητα ε, ε, γιατί το 2011 θα έρθει η πραγματική λιτότητα στα κράτη-μέλη. Αρχικά είχαμε πει το 2010, αλλά τελικά οι αποταμιεύσεις θα φανούν το 2011 ε, και ε, το κοινό και οι πολιτικές τάξεις όλων των χωρών θα πληγούν ακόμη περισσότερο το 2011. Αυτό είναι το γενικότερο πνεύμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να το παγώσουμε αυτό το πνεύμα της κρίσης για τα κομμάτια του προϋπολογισμού. Αφενός υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αφετέρου όμως Έχουμε ε, και ένα είδος ε, χρηματοπιστωτικής ειρήνης της Ευρώπης, δεδομένου του κλίματος χρειάζεται και αυτό. Πρέπει να αποφύγουμε ε, αυτό τον κατακαιρματισμό της Ευρώπης λόγω της ε, κρίσης, τον διχασμό της Ευρώπης λόγω της ε, κρίσης. Οφείλουμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στο κίνδυνο παγώματος των τμήματων του προϋπολογισμού λόγω μιας προσωρινής λιτότητας και αφετέρου να παράσχουμε στην Ευρώπη αυτή την οικονομική χρηματοπιστωτική ειρήνη για μια σειρά ετών, επιτρέποντας έτσι στην Ήπειρο να ενωθεί και να αντιμετωπίσει τις άλλες προκλήσεις που είναι πολυάριθμες και πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινέ απαντήσεις και μια τελευταία παρατήρηση θα κάνω ε, απαντώντας στον κύριο Κάλφιν, στον κύριο Φαν και σε εσά πρόεδρε. Ε, ε, δεν μειώνεται ο προϋπολογισμός, αυξάνεται. Κατά τι. Ε, αν δεν είχαμε τον ετήσιο προϋπολογισμό το 2011, θα έχουμε αύξηση. Δηλαδή με τα 12 ε, τιμόρια θα έχουμε ουσιαστικά ε, αύξηση σε σχέση με το 2010. Otherwise, we have a prognosis. Με τις προγνώσεις, ακόμη και με τη λιτότητα, Ε, παρά τη θέση του Συμβουλίου έχουμε μια αιωνία ανάπτυξη που προβλέπεται για το 2011 παρά τη λιτότητα ξαναλέω. Ε, η πιστός ανάπτυξη υποχρεώσεων πρέπει να κυμαίνονται στο 1,14 περίπου της 100 του ΑΕΠ για το 2011. Είναι ρεαλιστικό αυτό. Οι πληρωμές κατά τι θα υπερβούν το 1%. Δεν προδικάζω, δεν προεξοφλώ το, το, την έκβαση των ε, ετησίων διαπραγματεύσεων, αλλά και ακόμη και με το τωρινό κλίμα ε, διαβλέπουμε μία αύξηση, μία μικρή αύξηση αν υπάρχει συμφωνία για το προϋπολογισμό το 2011. Πρέπει επίσης να νόμιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός, όπως είπε και ο πρόεδρος Λαμασούρ, Πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό συνιστά τη θέμενη αξία. Ένα ευρώ που δαπανάται καλύτερα σε και επίπεδο ένωσης ε, από ότι σε εθνικό επίπεδο. Πώς ε, θα επιτύχουμε ένα συνδυασμό αυτών με ομαδοποίηση των πόρων προφανώς, με αντιμετωπίση ε, κοινών προκλήσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε, από τα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη απάντηση στι φυσικές καταστροφές, ένα ουσιαστικό ζήτημα που πλήττει την ε, ε, Ήπειρό μας και ε, νομιμοποίηση της αξιολόγησης της μη Ευρώπης ή της λιγότερης Ευρώπης. Και αυτό είναι μέρος των τωρινών διαπραγματεύσεων. Και ε, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει εξολόγηση της μη Ευρώπης ή της λιγότερης Ευρώπης. Ε, κατά τη γνώμη μου ε, θα ήταν αυτό ένα καλό έγγραφο υποβάθρου για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση. Βλέπω ότι έχουν τις αμφιβολίες τους τα μέλη της Επιτροπής. τέλος πάντων κατά τη γνώμη μου και από εδώ που κάθομαι εγώ στο Προεδρείο μου φαίνεται εφικτό αυτό. Εάν ε, ε, είναι να εκπονήσετε ένα πραγματικό έγγραφο, δεν μπορεί αυτό να γίνει γρήγορα Πάντω για τι διαπραγματεύσει για την περίοδο μετά το 2013 οφείλουμε να συνυπολογίσουμε και ε, το αρνητικό εναλλακτικό κόστος, ε, δηλαδή λιγότερη Ευρώπη και έλλειψη απαντήσεων στις ε, κοινέ προκλήσει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης. Αυτές τις παρατηρήσεις θα κάνω. Μετά με ρωτήσατε τι θα γίνει με το πακέτο, αν θα ενταχθεί. Μα πρέπει να κάνουμε επιλογή για τους ίδιους πόρους. Ε, είναι μια, ένας ουδέτερος ε, τελικός κατάλογος, ναι μεν, αλλά για το μέλλον πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Ε, ευχαριστώ. Εμείς σας κατευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, λέει ο Πρόεδρος. Δύο πράγματα κρατάω από αυτά που είπαμε σήμερα το πρωί. Πρώτον ότι στην Κομισιόν μαζί με 23 επίσημες γλώσσες υπάρχει και 24η σωματική τη αυτή για την οποία ίσως πρέπει να προσλάβουμε και σωματικούς διερμηνείς και διερμηνεύτριες. Δε, έπειτα βλέπω ότι, ότι γίνατε και εσείς τώρα. Γιατί αν περιοριστούμε σε αυτά που μας έλεγε ο Μέγας Βρετανός Πρωθυπουργός της Ισραήλ θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε. Έλεγε είμαι συντηρητικό για ό,τι λειτουργεί, αλλά όχι για ό,τι λέει λειτουργεί. Και ξέρουμε όλοι κύριε Επίτροπε ότι ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός δεν λειτουργεί. Χάρη όμως στις κοινέ μας προσπάθειες θα λειτουργήσει και έτσι θα γίνουμε όλοι τόροι. Θα συνοδεύσω μια στιγμή τον Επίτροπο. Η Αντιπρόεδρος θα προεδρεύσει όσο τον ξεπροβοδίζω Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ακόμη αρκετά πράγματα να κάνουμε και θα παρακαλούσα να συνεχίσουμε. Τώρα θα συζητήσουμε τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 10 και είμαι βέβαιος ότι ο Ράιμερ Μπέγκε και ο Λάσλο Σούριαν θέλουν επίσης να συζητήσουν το διορθωτικό προπολογισμό αριθμός 10 και τον το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 9 και παρακαλώ το Λάσλο να κάνει την εισαγωγή. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνοψίσουμε και τα δύο, δεν χρειάζεται δηλαδή το ένα να συζητηθεί ανεξάρτητα από το άλλο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Συμφωνώ με το, το σχέδιο του διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 9. Και όσον αφορά το διορθωτικό προπολογισμό αριθμός 10, αυτό θέλει λίγο περισσότερη συζήτηση. Αλλά ξεκινώντας από το τέρμα, από το τέλος ζητώ από την Επιτροπή να το στηρίξει. Έχω όμως δύο ή τρεις επιφυλάξεις. Ε, η πρώτη είναι ότι πρέπει να πιέσουμε την Επιτροπή να βρει άλλες λύσεις, όπως η μείωση των γραμμών ως προβλέπονται στο διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 10 το, η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι αυτή, αυτός ο διορθωτικός υπολογισμός αριθμός 10 δεν μπορεί να κριθεί από μόνο του. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε τις 53 αν θυμάμαι καλά γενικές μεταφορές και εν ώψη των γενικών μεταφορών θα αποκομίσουμε και μία ιδέα για την πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011. Δηλαδή, ε, σκέφτομαι ε, να εξετάσουμε το 1β, ε, το κεφάλαιο 1β, διότι η Επιτροπή αυξάνει κατά πέραν του ενός δισεκατομμυρίου αποδεικνύοντας σαφώς ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου και του εισηγητή σας πέρυσι ε, ε, δεν ε, απέδωσαν και τώρα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να καλύψουν ε, το, τη διαφορά μεταξύ ε, της δεσμεύσεως και της πληρωμής. Άρα η μεταφορά του ενός δισεκατομμυρίου αποτελεί ε, μία φιλοφρόνηση προς το μέρος μας. Συγχρόνως όμως θέλουν να μειώσουν το κεφάλαιο 1β ε, για τον προϋπολογισμό του χρόνου. Θέλω λοιπόν να δηλώσω και πάλι ότι ε, θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό θα αλλάξει μέσα στο χρόνο. Τώρα όμως δεν συζητάμε τον προϋπολογισμό του 2011, απλώς το αναφέρω διότι το θέμα αυτό συνδέεται με το προηγούμενο. Και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Δεν ζητώ να υπάρξει μία συνεδρίαση συγκεκρισμένων των θυρών, αλλά αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ένα τεχνικό θέμα. Δηλαδή, σε περίπτωση όπου δεν υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο για τον προπολογισμό του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί για κάποιους μήνες να ζήσει με τα 12 τετιμόρια. Δεν νομίζω ότι θα είναι μία διαδικασία που θα κρατήσει ένα χρόνο, αλλά σίγουρα ορισμένους μήνες και αφού ο τροποποιηθεί ο προπολογισμό του 2010 θα μειωθεί το ποσό κατά ένα δισεκατομμύριο και πέρυσι με τη στήριξη και χθε με τη στήριξή σας είπα στον τριμερή διάλογο ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να στηρίξει τον διορθωτικό προπολογισμό αριθμό 10 μόλις συμφωνήσουμε. Δηλαδή υπάρχει μία υποαίρεση ε, ε, ε, συμφωνία της Επιτροπής αυτής. Βεβαίως ελπίζω ότι θα υπάρξει μία συμφωνία τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο κάποια στιγμή αλλά ιδεοδός πριν την 1η Ιανουαρίου καλό θα ήταν ε, να, έχουμε, να περάσουμε την τελευταία μέρα του χρόνου μαζί στο Στρασβούργο παραδείγματος χάρη αλλά ουσιαστικά το βασικό θέμα είναι ο διορθωτικός προπολογισμό αριθμός 10. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος κυρία Χάουγκ. Βεβαίως στις 3 το απόγευμα όταν θα έχουμε την συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση αλλά πρέπει να το μεταφέρουμε στην Επιτροπή στην 1η Δεκεμβρίου οπότε ελπίζουμε ότι θα έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο οπότε τα πράγματα θα προχωρήσουν εκ του παραλίλου δηλαδή πρώτα συμφωνία με το Συμβούλιο και μετά διορθωτικός προπολογισμό αριθμών 10. Ο κύριος Φέρμ. Αν πρόκειται να συζητήσουμε με το απόγευμα, θα περιμένω στο απόγευμα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει κάτι να συζητήσει επ' αυτού. Όχι, δεν βλέπω. Τώρα, σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμός 9, δεν ακούσαμε καμία διαμαρτυρία όταν ο εισηγητής είπε ότι θέλει να την υιοθετήσει ως έχει και έτσι ερχόμαστε τώρα στο σημείο της ημερησίας διατάξεως 8 και εδώ θα έπρεπε να κινητοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης το οποίο είναι υπόθεση του Ράιμερ Βέγγε, στον οποίο δίνω το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι αρκετά σύντομος. Εδώ πρόκειται στην για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την καταστροφή στην Πορτογαλία, στη Μαδέρα το 2010 και δεύτερον για την ε, ε, ε, ε, τις καταστροφές που προκάλεσε η καταιγίδα Ξύνθια ή στη Γαλλία πάλι το 2010. Οι πορτογαλικές αρχές ε, είχαν αξιολογήσει το σύνολο των ζημιών σε 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ που είναι 1,6 του πορτογαλικού ΑΕΠ και άρα έχει ξεπεραστεί το κατόφλι των 0,6% του ΑΕΠ σύμφωνα με τον κανονισμό της κινητοποίησης του Ταμείου Ελληνικής για μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές άρα και η Μαδέρα εμπίπτει στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Όσον αφορά στην Γαλλία υπολογίζουμε περίπου 1,4 δις στην περίπτωση αυτή πρόκειται για αριθμούς οι οποίοι βρίσκονται ε, κάτω από το σύνηθες κατόφλι και γι' αυτό ε, η ε, Επιτροπή έλεγξε την περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτακτου κανονισμού στο σημείο 2.2 και εφόσον πρόκειται για έκτακτη καταστροφή θα πρέπει να να αξιολογήσει κανείς ότι επηρεάστηκε η ζωή των κατοίκων της περιοχής, η βιομηχανική ανάπτυξη και η σταθερότης. Λοιπόν, 2,5 ε, εκατομμύρια για την ε, ε, Πορτογαλία και για την Γαλλία σύνολο 66 εκατομμύρια προβλέπεται ότι η ψηφοφορία επί του θέματος θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου στην Επιτροπή το Δεκέμβριο εις το, στην Ολομέλεια και όσον αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 9 ε, εφόσον υπάρχει το πρόγραμμα ανακάμψεως και ιδίως ε, το πρόγραμμα των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας έχουμε ένα πρόγραμμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιληφθεί ότι στο πρόγραμμα ανάκαμψης θα πρέπει να καλυφθούν πλήρως και αυτές οι απαιτήσει και το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμά της επί του θέματος και παρακαλώ να το πράξει. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Και πάλι για όλους τους συναδέλφους, διότι ε, συμπεριλαμβάνεται και ο Ανδρέα. Ε, η προθεσμία είναι 10 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι, δηλαδή αύριο το μεσημέρι και έχετε μέχρι τότε τη δυνατότητα να υποβάλλετε μία τροπολογία. Στην αρχή ήταν 12 του μηνός, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Ο Μιγγέλ Πόρτας είχε ζητήσει το λόγο. Κοιτάξτε. Ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Είναι προφανές ότι είμαι υπέρ της κινητοποίησης αυτού του ταμείου. Θα ήθελα παρόλα αυτά να προτείνω το εξής, να τροφοδοτήσω τη συζήτηση αν θέλετε. Οι πλημμύρες ε, στη Μαδερά έλαβαν χώρα το Φεβρουάριο. Πέρασαν 8 μήνες. Τα κονδύλια που τόσοι ή δεν είναι υψηλά, 31 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, για ζημιές ε, που εκτιμώνται σε 1,8 δις. Οπότε είναι μικρή υποστήριξη από πλευράς της Ένωσης. Επίσης έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η βοήθεια και θέλουμε να αναρωτηθούμε για το μηχανισμό βοήθειας. Φτάνει Φτάνει χειμώνα σιγά σιγά στη Μαδέρα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη και ε, εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσκολίες ε, ε, του πορτογαλικού κράτους και των περιφερειών οικονομικές δυσκολίες. Πολλές οικογένειες ε, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ε, διότι ε, δεν έγιναν τα απαραίτητα έργα για τις κοίτες των ποταμών, για τις κατολιστήσεις. Θυμάστε τι έγινε το Φεβρουάριο, υπήρχαν σοβαρές ζημιές μετά τις πλημμύρες. Οπότε θα θέλαμε αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης να είναι πιο ευέλικτο. Όταν ε, κυρίως ε, ε, διερχόμεθα μια περίοδο λιτότητας και θέλουμε να δαπανούμε τα ελάχιστα δυνατά κονδύλια κάνοντας πολλά πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τον Απρίλιο μια μικρή αντιπροσωπεία του ΕΛΚ πήγε στη Μαδέρα στην περιφέρεια ακριβώς που είχε πληγεί από τις πλημμύρες ήταν εκεί ο κύριος Γκαρίγκα, ο κύριος Φερνάντες, ο κύριος Καρβάλιο και εγώ. Και μας δέχτηκε η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί Μείναμε δύο μέρες εκεί, συναντήσαμε πολλούς, κάναμε συνεντεύξεις τύπου και εξηγήσαμε ότι η Ένωση και το Κοινοβούλιο θα σταθούν στο πλευρό της περιφέρειας αυτής που είχε υποστεί τέτοια καταστροφή. Όταν πήγαμε εκεί ήταν ακόμη αποδογυρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους, σπίτια χωρίς στέγη παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπίσουν το καλοκαίρι κανονικά. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς όπως έγινε και για την περιοχή των λιμνών στην Ιταλία και για την Ακούιλα. το ίδιο να γίνει και για την Πορτοκαλία, την σασόρες και τη Ματέρα. Ναι, νομίζω ότι επανακάμπτει και πάλι το πρόβλημα σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης ότι περνάει τόσος χρόνος μεταξύ του γεγονότος που προκάλεσε τη ζημιά και την διάθεση της πιστώσεως και των κεφαλαίων. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα μεταξύ των δύο αυτών σημείων. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να επιταχύνουμε. Ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί πόσο μπορούν να ε, βραχύνουν τα, τις ε, διοικητικές διαδικασίες. Δηλαδή θα πρέπει ε, να αξιολογήσουν πιο γρήγορα και να υποβάλουν την αίτηση γιατί αυτό διαρκεί αρκετά, αρκετό χρόνο χρόνο αλλά ήδη να βρισκόμαστε στον Νοέμβριο από τον Ιανουάριο είναι αρκετός χρόνος. Ο Σαλβαντόρ. Πρέπει να πούμε ότι έχουν επιταχυνθεί διαδικασίες. Ίσως θυμάστε τον κικαιώνα της Σλοβακίας όταν υπήρξαν οι καταστροφές στη Σλοβακία. Χρειάστηκε ένας χρόνος ενώ εδώ μιλάμε για πλημμύρες του Φεβρουαρίου, είμαστε τον Νοέμβριο και όντως Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία και οι αρχές θα πληρωθούν όταν ε, παρεμβαίνουν πολλές ε, διοικήσεις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές χρειάζεται χρόνο. Το πιο μακρύ ε, σημείο είναι η κοινοτική διαδικασία διότι κινητοποιήσαμε γρήγορα το Ταμείο, αμέσως συμφωνήσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες, άρα το ουσιαστικό πρόβλημα είναι η διασύνδεση μεταξύ της εθνικής αρχής με ε, την κοινοτική αρχή. Πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση των ζημιών, επιλογή ε, των ε, διορθωτικών μέτρων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά όταν καταφέρνουμε να μειώσουμε το χρόνο κάτω της χρονιάς, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό. Ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι αυτές οι διαδικασίες και όλες οι διαδικασίες ε, που ε, σχετίζονται με φυσικές καταστροφές ε, πρέπει να βελτιστοποιηθούν, να είναι ταχύτατοι μηχανισμοί. Παρόλα αυτά, στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρα άρχισαν αμέσως τα έργα. Δεν μπορούμε παρά να το καταγράψουμε αυτό. Την ταχύτητα με την οποία η, περιφερειακή, η τοπική αυτοδιοίκηση της Μαδέρα προχώρησε στα έργα παρότι περιμένει ακόμη τα κονδύλια και από την Ένωση και από ε, την κυβέρνηση. Τα κονδύλια δηλαδή που έχει υποσχεθεί η Πορτογαλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες ε, προς απόφαση. Θα ψηφίσουμε 18 Νοεμβρίου και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο οπότε θα μπορέσουν ίσως να μεταβιβαστούν τα χρήματα στην Πορτογαλία πριν τελειώσει ο χρόνος. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα ή μάλλον στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την κινητοποίηση του ο, Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση όπου υπάρχουν δύο θέματα που δεν πρέπει να αποφεστούν σήμερα αλλά πρέπει να συζητηθούν. Και η Μπάρμπαρα έχει το λόγο για τα σημεία 9 και 10 της ημερησίας διατάξεως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, έχει, στο Ταμείο έχει υποβληθεί ένα γερμανικό αίτημα για 1150 εργαζόμενους από τέσσερα εργοστάσια στη Βάδη Βιρτεμβέργη. Στον τομέα της πρέσας. 8 εκατομμύρια και κάτι ευρώ έχουν ζητηθεί από τη Σλοβενία για να βοηθηθούν 1544 απολυόμενοι στον τομέα της ένδυσης και 2.250.000 περίπου, περίπου συνολικά. Η υποβολή τροπολογιών λήγει στις 12 Νοεμβρίου και η, ψηφοφορία θα γίνει 18 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας. Πριν όμως από αυτό θα ήθελα να επανέλθω στις ψηφοφορίες που θα κάνουμε σε λίγο. Έξι αιτήματα κινητοποίησης χρήσης αυτού του ταμείου από την Ολλανδία. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ψηφίσουμε σε λίγο. Έχει υποβληθεί μία τροπολογία του κυρίου Αλβάρο και Όκλαντ. Των κυρίων Αλβάρο και Όκλαντ. Είμαι υπέρ της τροπολογίας αυτής που ζητάει περισσότερες πληροφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον τρόπο χρήσης αυτών των ποσών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ταμείο στοχεύει ακριβώς την υποβοήθηση των εργαζομένων για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας με συμβόλαια περιορισμένου χρόνου. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σε όσους συντάσσουν τροπολογίες ότι για την αναθεώρηση της λειτουργίας του Ταμείου αυτού οι προτάσεις συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση πόρτας για τη χρηματοδότηση και λειτουργία, επαναλαμβάνω, του Ταμείου αυτού προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Δεν περιμένουμε δηλαδή να μας κάνει προτάσεις η Κομισιόν για την αναθεώρηση του Ταμείου, απλώς βλέπουμε αν πληρούνται οι στόχοι που ζητούν να πληρούνται οι διάφοροι συνάδελφοι. Η κυρία Βέρτμαν. Η κυρία Βέρτμαν, θέλω να αναφερθώ στην περίπτωση Heidelberg και Druckmaschinen, διότι ε, είναι μια διεθνής επιχείρηση και μπορώ να πω ότι είναι ένας πυλώνας των γερμανικών, της γερμανικής βιομηχανίας μηχανημάτων και βλέπω ότι υπάρχει μία αίτηση από αυτήν την ε, ε, ε, επιχείρηση και πρέπει να σας πω ότι το 5-206 είχαν 220 εκατομμύρια μέχρι την επόμενη χρόνια 300 μετά 390 και μετά 370 εκατομμύρια δηλαδή ε, τώρα βλέπουμε ότι πλέον η επιχείρηση ε, έχει ζημιές αλλά ε, αυτή τη στιγμή ανακάμπτει. Πρέπει λοιπόν να δούμε διάφορες αναφορές ή στον τύπο για το 2006 διότι τότε η επιχείρηση αυτή κατήρτησε μία επιχείρηση στην Σαγκάλα Σανγκάη ε, και συμμετείχε με μεγάλες ζημιές. Δηλαδή ε, ήδη το 2006 ε, η αγορά της Κίνας ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για αυτή την επιχείρηση. Βεβαίως καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτή η επιχείρηση για να μπορεί να θέτει το αίτημά της. Αλλά αυτό που εμένα με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι ότι ακόμη και αν υπάρχει ανάκαμψη η Γερμανία είναι ε, μια χώρα η οποία έχει ε, ε, υψηλά ημερομίσθια και υπάρχουν απολύσει 1.100 εργαζομένους αλλά στις ασιατικές χώρες υπάρχουν αυξήσεις προσωπικού ε, σαν Αυστριακή λοιπόν βλέπω ότι διαβάζω στον γερμανικό τύπο πω ότι με ευρωπαϊκά χρήματα στηρίζουμε το, την αγορά εργασίας του τρίτου κόσμου. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό να μειώνουμε το προσωπικό στην Ευρώπη, να στηρίζουμε με τα ευρωπαϊκά ταμεία και στην Ασία να αυξάνουμε το προσωπικό. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές και πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και προηγουμένως να συνυπολογιστεί και βεβαίως να υπάρξουν και περιορισμοί διότι βεβαίως ενδέχεται ε, να χρειαστεί να συζητήσουμε και για μια αμερικανική επιχείρηση που έχει θηγατρική στην Αυστρία, περιμένω ακόμη τους αριθμούς. Πρέπει όμως νομίζω να εξετάσουμε τους αριθμούς διαμέσου των ετών και εγώ εχθές το βράδυ έκατσα και κοίταξα αυτή την πορεία λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Ευχαριστώ κυρία Βέρτμαν. Όσον αφορά την επιχείρηση αυτή Heidelberger Druckmaschinen έχω προσωπική επαφή ε, μη με παρανοήσετε αλλά ξέρω ε, ε, γιατί η δικιά μου περιφέρεια είχε ζητήσει να εγκατασταθεί εις ε, την περιοχή μας αυτή η επιχείρηση διότι είμαστε μια περιοχή η οποία έχει ε, πληγεί από τη μείωση των ε, ορυχείων και είδατε όμως ότι έπρεπε αντί για μια περιοχή του, του χώρου 2 να πάει στην, σε περιοχή του χώρου 1 στις, σε, μία από τις, ε, σε ένα από τα πέντε κρατήδια τα νέα της, της ε, γερμανικής ε, επικράτειας και πρέπει να σας πω ότι δεν βοηθάμε μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες απολύουν αλλά βοηθούμε και τους απολυμένους οι οποίοι πλήττονται για να μπορέσουν και πάλι να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Με περισσότερες δεξιότητες, με καλύτερη εκπαίδευση θα επισέλθουμε στις λεπτομέρειες αυτές. Αλλά βλέπω τώρα ζητά το λόγο ο Λάσλο Σούριαν και ο Μίγκελ Πόρτας. Ε, ακριβώς αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή να είναι σαφές ότι τα χρήματα αυτά που στέλνουμε στους ετούντες δεν θα πάνε στην εταιρεία. Τέλος πάντων. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε λιγάκι. Διότι αν πάρω ένα άλλο παράδειγμα ας πούμε στο Ταμείο Αλληλεγγύης φάνηκε ότι υπήρχε κάποιος υπεύθυνο, όποτε υπάρχει υπεύθυνο για κάποια καταστροφή τότε πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα στην Κομισιόν. Στο μέλλον, όταν μιλάμε για το μέλλον του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, θα έπρεπε και αυτό το σημείο, αυτή τη ρήτρα να τη βάλουμε. Αν δηλαδή αποφασίσει ελεύθερα η εταιρεία ότι θέλει να μετεγκατασταθεί αλλού όπου είναι χαμηλότερη μισθή κτλ. Ζητούν λοιπόν αύξηση του κέρδους τους, τότε δεν ε, πρέπει να είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση. Γιατί η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι μεν εθνικό καθήκον, αλλά σε μερικές περιπτώσεις ενέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. και ένας λόγος που πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και για τον οποίο υπάρχει το ταμείο αυτό είναι για να βελτιωθεί και η εικόνα της Ένωσης. Αν συμμετέχει στο προ, στη δημιουργία του προβλήματος η εταιρεία τότε να πληρώνει και εκείνη. Δεν είναι καταλληλότερη στιγμή τώρα να το αποφασίσουμε αυτά αλλά τέτοιου είδους συζητήσεις πρέπει να γίνουν κάποτε. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που ακούσαμε. Μιγγέλ. Ε, ήθελα μία παρατήρηση να κάνω μόνο για αυτό το δίλημα που ετέθη από τη συνάδελφο. Είναι λογικό να προβληματιστούμε γι' αυτό. Ποιο είναι αυτό. Το... Η Γιούτα δίκιο έχει. Δηλαδή ε, υποστηρίζουμε τους ε, απολυμμένους και όχι την εταιρεία με αυτό το ταμείο. Από αυτή την πλευρά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρόταση που είναι σωστή, η πρόταση που λάβαμε. Τώρα, τι συμβαίνει. Αυτή η κατάσταση στην οποία μια πολυεθνική απολύει κάποιους και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης αλλού και μέσα στην Ευρώπη. Έτσι έχει συμβεί αυτό σε προηγούμενες, σε προηγούμενες αιτήσει. Ε, απολύονται στην Ιρλανδία και ανοίγει καινούργιο υποκατάστημα στην ε, Πολωνία. Ε, δεν συμβαίνει πρώτη φορά αυτό. Το Ταμείο δεν μπορεί να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ με τον Σούριαν. Θα χρειαζόμασταν ίσως, είπε, να έχουμε ένα άλλο μέσο, έναν άλλο κανονισμό που να εγγυάται ότι η Ευρώπη ε, θα υποβοηθεί από τα ταμεία όταν στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι έμεση χρηματοδότηση της μαζικής απόλυσης, δηλαδή έμεση χρηματοδότηση των μαζικών απολύσεων. Αυτό νομίζω είναι μια πραγματικότητα και δεν χρειάζεται να ε, ε, καλύπτουμε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η κυρία Βέρτμαν και πάλι και πάλι η κυρία Βέρτμαν. Ήθελα να διευκρινίσω τη θέση μου. Η θέση μου προς ε, το ε, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης σημαίνει ότι βεβαίως χαιρετίζουμε τις κινήσεις αυτές, αλλά είναι προφανές ότι όταν μία επιχείρηση απολύει είναι απολύονται οι ε, Ευρωπαίοι, οι κοινοτικοί οι οποίοι στηρίζονται αλλά ε, εάν ε, αυξάνει τις προσλήψεις σε ένα άλλο σημείο σημαίνει ότι υπάρχει κακή χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων και δημιουργούμε ένα φραγμό. Πρέπει να μην, ε, να μην πηγαίνει, ε, να μην κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί η εταιρεία αυτή ε, είναι σε ανθυρή κατάσταση. Πάει πολύ καλά. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Σας καταλαβαίνω. Ας μην κάνουμε συζήτηση όμως τώρα. Διότι διότι αν ακολουθήσουμε αυτό και πούμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση, τότε ε, θα είμαστε αντίθετοι σε αυτό το οποίο ε, είχαμε ε, καταψηφίσει πριν από 20 χρόνια, δηλαδή την προγραμματισμένη οικονομία. Κάνουμε ορισμένες επιλογές είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, σας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά ο Αλεξάνδρ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Όσο δύσκολο και να είναι το θέμα της Heidelberg και Druck, εάν δεν υπήρχε η στήριξη θα είχε πτωχεύσει η εταιρεία αυτή. Και αυτό αποδεικνύουν οι αριθμοί και δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας αν επιβιώνει η εταιρεία ή όχι διότι όπως είπε και η Γιούτα τότε θα εφαρμόζουμε μία προγραμματισμένη οικονομική πολιτική αλλά ε, υπάρχει και η Νόκια όπου υπήρξε μετακίνηση μέσα στην Ευρώπη από τον Μπόχουμ στη Ρουμανία Υπάρχει το Ταμείο Προσαρμογής το οποίο εμπλέκεται όχι πάντοτε πολύ σαφώς παραδείγματο χάρη το είδαμε και στην περίπτωση της Νόκια αλλά η ερώτησή μου στη Heidelberger Druck είναι ότι αν υπάρχει η απόλυση η οποία δεν ευθύνεται στην παγκοσμιοποίηση γιατί δεν έχει παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που θα ήταν η σωστή λύση διότι εάν περνούμε από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπάρχει ίσως μία κατάχρηση του Ταμείου αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι γίνεται, τι στηρίζεται από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και αν χρειαζόταν να εμπλακεί άλλο ταμείο, ε, αν στην δηλαδή έπρεπε να εμπλακεί το κοινωνικό ταμείο, τότε γιατί χρηματοδοτούμε μέσω του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Γιατί νομίζω ότι στην Heidelberger Druck ο σωστός, η σωστή πηγή για τη χρηματοδότηση έπρεπε να είναι το κοινωνικό ταμείο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, κατάλαβαν ε, οι ενδιαφερόμενοι ότι μπορούν να καλυφθούν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Τα ίδια λέμε συνέχεια. Όποτε μιλάμε για συγκεκριμένες προτάσεις χρήσης του Ευρωπαϊκού Αυτού Ταμείου. Θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται για ένα μέσο ή εργαλείο που διαστρεβλώνει την αγορά Άκουσε Γιούτα. Με όλο το σεβασμό που σου οφείλω διαφωνώ. Ο διαχωρισμός μεταξύ επιχορηγήσεων, το κατά πόσο επιχορηγήσεις πηγαίνουν στις επιχειρήσεις τους εργαζόμενους είναι κάτι το λανθασμένο διότι πολλοί προβλέπουν ήδη στην λειτουργία της επιχείρησής τους ότι θα χορηγηθούν τέτοιες επιχορηγήσεις και πολλές φορές εποφελούνται και για να απολύσουν. Έμεσα λοιπόν την επιχείρηση βοηθούν πάντοτε. Ο Λάσλο επίσης είπε κάτι πολύ σωστό. Είναι αδύνατον είπε να γνωρίζουμε κατά πόσον το ταμείο αυτό προκάλεσε την απόφαση με την κατάσταση της επιχείρησης, σε τι βαθμό. Και όσους όρους και να βάλουμε, πάντοτε θα υπάρχουν επιχειρήσεις που θα κάνουν κατάχρηση του ταμείου αυτού. Το όλο θέμα λοιπόν στρεβλώνει την αγορά. Όσο γρηγορότερα το καταργήσουμε αυτό το ταμείο, τόσο το καλύτερο θα είναι για το μέλλον αν θέλουμε τουλάχιστον να αποφύγουμε την παλιότερη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο Σαλβαδόρ. Και εγώ με όλο το σεβασμό που οφείλω στον κύριο Μποκρός θα έπρεπε να του πω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του ταμείου αυτού είναι ότι ακριβώς δεν δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Είναι το μόνο μέσο που διαθέτουμε που απευθύνεται κατευθείαν στον εργαζόμενο. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν προέρχεται, βασίζεται στις δημοσιονομικές προοπτικές, στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές που το είχαν ιδρύσει ως ανταπόκριση, ad hoc ανταπόκριση της Ένωσης σε έκτακτες καταστάσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι ορισμένων επιχειρήσεων πλήττονταν από την παγκοσμιοποίηση. Και στη συνέχεια λόγω της κρίσης δόθηκαν και άλλες δυνατότητες παρέμβασης στο Ταμείο αυτό και όλες οι επιχειρήσεις που λόγω της οικονομικής κατάστασης γενικότερα μπορούσαν να τεθούν εν κινδύνο, είχαν το δικαίωμα να υποφεληθούν. Πολλές απευθύνθηκαν στο Ταμείο. Αρκεί να διαβάσετε την ανάλυση που έκανε ο Πόρτας για την ιστορία του Ταμείου και θα δείτε ότι ο αριθμός των ετοιμάτων αυξήθηκε εκθετικά τα τελευταία χρόνια όχι τόσο λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλά μάλλον λόγω της οικονομικής κρίσης. Η κατάσταση λοιπόν αυτή έχει χαρακτήρα όλος εξαιρετικών. Και αυτό θα περιοριστεί χρονικά, μέχρι το 2011, είπαμε. Και όταν επανέλθουμε στην παλαιότερη, στην αρχική κατάσταση δηλαδή τότε, τότε λέγω δεν θα υπάρχουν πια τέτοια προβλήματα όπως η κατάσταση για την οποία μιλήσαμε. Τελικά νομίζω ότι το ταμείο αυτό είναι πολύ χρήσιμο και κάνει πιο ορατή την ένωση μεταξύ των εργαζομένων. Είναι το μόνο εργαλείο και μέσο, επαναλαμβάνω, που επιτρέπει μία πρακτική και συγκεκριμένη βοήθεια για τους εργαζόμενους. Εκτός βέβαια αν στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές από το 2013 και μετά καταφέρουμε να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία του κοινωνικού ταμείου. Αλλιώς και μέχρι στιγμής μόνο αυτά τα δύο ταμεία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπω άλλο να ζητά το λόγο, οπότε η Μπάρμπαρα μπορεί να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα να καταλήξω σε συμπεράσματα, διότι όπως ε, πολλοί ε, σωστά εξήγησε και ο Σαλβαντόρ, ε, το ταμείο αυτό αποσκοπεί στην, στο να βοηθά τους εργαζομένους και όχι την επιχείρηση. Θέλω να καθησυχάσω την κυρία Βίτμαν. Ε. Δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ε, Κινέζους εργαζομένους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Ταμείου. Ε, ο στόχος του Ταμείου είναι να ε, παράσχει στήριξη στους εργαζομένους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα κονδύλια θα μπουν στις τσέπες των δικαιούχων των εργαζομένων που χάρη σε αυτά θα διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες θα μπορέσουν να καταρτιστούν επαγγελματικά Πέρα από τα μαθήματα γλώσσες, μιλάμε για ε, τεχνική επαγγελματική κατάρτιση. Είναι πραγματικά ε, σημαντικό ε, αυτό το ταμείο και θα πρέπει να εξετάσουμε με πάσα σοβαρότητα την χρήση των κονδυλίων του ταμείου και όπως ζητάει και ο κύριος Άλβαρο μέσα στην τροπολογία του θα εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα της χρήσης των κονδυλίων του ταμείου. Βέβαια, η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ε, κρατών μελών έχουν δίκιο. Υπάρχει ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, της τάξης του 35%. Δηλαδή κάθε εθνική κυβέρνηση ελέγχει την ε, χρήση αυτού του ταμείου και φυσικά δεν είναι ανόητοι όσοι διαχειρίζονται τα κονδύλια του ταμείου. Είναι χρήσιμη πάντως η συζήτηση που γίνεται ίσως η Επιτροπή να τοποθετηθεί διαφορετικά για το Ταμείο προσαρμογή στην ε, Παγκοσμιοποίηση. Το Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα διαφορετικό ταμείο αυτή τη φορά. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά το 2013 πρέπει να επιβιώσει, να παγιωθεί το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσει η συζήτηση αυτή. Η προθεσμία για τροπολογίες για τις δύο εκθέσεις της Βάρβαρα Ματέρα είναι 12 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί. δηλαδή διαφορετικά από ό,τι είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης του Ράινερ Μπέγκε. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης και πρόκειται ε, για τη χορήγηση εγγύσεων και ο Ιβάιλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε εκτεταμένα συζητήσει αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Τι έγινε στο ενδιάμεσο διάστημα. Ήδη ε, ε οι τροπολογίες ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που αφιέρωσαν κάποιο από το χρόνο τους για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Από τις τροπολογίες νομίζω προκύπτει ότι εντοπίσαμε διάφορες ε, βασικούς τομείς παρουσιάζουν ενδιαφέρον ε, δημοσίευση των εργασιών, κοινοποίηση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μεταξύ άλλων. Αυτή είναι η γενική ιδέα της έκθεσης, με να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις νέες απαιτήσει που τώρα ζητούμε από την Τράπεζα και την ενίσχυση της ίδιας της δομής της ισχύω ε, της ε, τράπεζας. Μία δεύτερη κατηγορία τροπολογιών σχετίζεται με το πεδίο της ε, εντολής της τράπεζας. Κάποιες τροπολογίες συγκεκριμένα ζητούν ενεργότερες δράσεις για τη μείωση της στόχης για το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Και πάλι ε, ε, αυτό είναι σημαντικό το ζήτημα και πρέπει να βρούμε την ε, κατάλληλη διατύπωση διατηρώντας άθικτο το ρόλο, το προφίλ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτό είναι το γενικό πνεύμα που διαπνέει τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Δεν θέλουμε να τροποποιήσουμε την ταυτότητα της τράπεζας, θέλουμε να ενισχύσουμε τα δυνατά της σημεία περαιτέρω. Τρίτον, συγκρότηση ενό ε, μηχανισμού εποπτείας παρακολούθησης αναθεώρηση ε, των τρεχουσών πρακτικών. Ποιο είναι ο ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων των λοιπόν ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διεθνού εμβέλεια. Αυτό είναι ένα νέο σημαντικό στοιχείο για τις απαιτήσει που προβάλλουμε στην τράπεζα. Νομίζω ότι όλοι ακολουθούμε την ίδια ρότα και πρέπει να επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο τη διατύπωση για να καταλήξουμε στην τελική διατύπωση. Ακόμη αναμένουμε προτάσεις από όλες τις ε, συναρμόδιες επιτροπές. Σήμερα ε, ψηφίζουν στην Επιτροπή Ανάπτυξης, είναι η τελευταία επιτροπή που ψηφίζει σήμερα για τις τροπολογίες. Θα έρθω σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές ε, αμέσως μετά την ψηφοφορία για να δούμε, να αναθεωρήσουμε τους καταλόγους ψηφοφορίας και να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι σκιώδης για το ΕΛΚ και συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις του κύριου εισηγητή, ιδιαίτερα ως προς τις τροπολογίες. Τρεις υποβλήθηκαν. Τρεις υποβάλαμε μάλλον και ακολουθήσαμε την εξή στρατηγική. Πρώτον, τις, ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι οι επενδύσεις προφανώς, έχει αυτονομία, συλλέγει κεφάλαια και δεν μπορεί να δαπανά χρήματα εκτός ένωσης. Ούτε έχει το δικαίωμα να ρισκάρει χρήματα εκτός ένωσης. Δεύτερον, όπως υπόθηκε πολλές φορές, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια των προοπτικών της Λισαβόνας. Οι τροπολογίες μας λοιπόν δύο, σε δύο στοιχεία βασίζονται. Πρώτον, να καθοριστεί σαφέστερα ο ρόλος της ΕΤΕ ως προς την συμβολή της στην ανάπτυξη στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχουν 10-12 χώρες με τις οποίες έχει συμφωνίες η Ένωση. Είναι φυσικό λοιπόν η Ευρώπη να παρακολουθεί τη δράση της ΕΤΕ εφόσον έχει εγγύηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τον οποίο μιλήσαμε πριν. 10% σας θυμίζω των επενδύσεών της την εγγυήσεων και κατά 16, δισεκατομμύρια καλύπτονται αυτές οι εγγυήσεις. Οι τροπολογίες μας λοιπόν προτείνουν τρόπους ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι βέβαια αναπτυξιακή τράπεζα αντίθετα με την παγκόσμια και άλλους δημοσιονομικούς οργανισμούς και το κεφάλαιό της ανήκει στην Ένωση. Επομένως πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί η σταθερότητά της και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι να μην κάνει επενδύσεις δηλαδή παρακινδυνευμένες. Δεύτερον, δεύτερη τροπολογία, ο προϋπολογισμός της Ένωσης και οι δυσκολίες έγκρισής του. Αντί να αυξήσουμε τα ποσά για κάθε περιφέρεια προτείναμε να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο επαναχρησιμοποίησης των πόρων μεταξύ περιφερειών. Δεν ζητήσαμε πρόσθετο ποσά. Ζητούμε τη μετακίνηση, τη μεταφορά κεφαλαίων σε προς όφελος των περιφερειών που θα αποτελέσουν προτεραιότητα σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει για την εξωτερική πολιτική και άλλους τομείς. Τρίτον, να ενισχυθεί ο δημοσιονομικός έλεγχος μέσω ενός νέου εργαλείου συνεργασίας με περισσότερη, περισσότερο συντονισμό των αρμοδίων αρχών για τον προϋπολογισμό που από κοινού θα αποφασίσουν πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο όργανο ή μέσο. Όλα αυτά βασίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Άλλη τροπολογία. Ο έλεγχος που γίνεται για τα δημοσιονομικά προγράμματα της ΕΤΕ για εξωτερικές δράσεις και για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ανάπτυξης ζητούμε να υπάρξει μια μεγαλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ των παραγόντων που λαμβάνουν τις αποφάσεις και τρίτον να αυξηθεί το περιθώριο αναχρησιμοποίησης των πόρων μεταξύ των περιφερειών για να υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος χωρίς να επιβαρύνεται ο υπολογισμός. Ευχαριστώ κύριο Στόγεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήμουν σκιώδης εισηγήτες για την γνωμοδότηση στην ΕΚΟΝ και μπορώ να σας πω ότι συνεργαστήκαμε με τον εισηγητή και ότι είναι μια σωστή εργασία αυτή την οποία εξετάζουμε σήμερα. Πρέπει όμως να συνεχιστεί η συνεργασία διότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένες ακαμψίες ε, οι οποίες ε, ε, εντείνονται από ορισμένες τροπολογίες όπως η τροπολογία 21 η οποία προτείνει στην ε, Διεθνή Τράπεζα η οι ε, ε, εγγυήσει να μπορούν να να αιτιολογούνται ε, προς όφελος των εργαζομένων. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να βάζουμε τέτοιους περιορισμού, αλλά θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ε, όπως ε, είπε ο εισηγητής ευχαρίστως θα συζητήσει με τους άλλους εισηγητές οπότε ε, του ξαναδίνω το λόγο τώρα για να καταλήξει. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική για όλους διατύπωση, γιατί σκεφτόμαστε πάνω κατά τα ίδια πράγματα, αλλά θυμίζω ότι είμαστε και σε διαδικασία συναπόφασης. Χρειαζόμαστε την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Επίση, και νομίζω ότι από πλευρά του Κοινοβουλίου θα έχουμε δυσκολίε να πείσουμε το Συμβούλιο, όπω είπε και ο κύριος Κόλλιν, για την αύξηση των ορίων ή την αύξηση τη ευελιξία με, με τις υφιστάμενε οροφές, τα υφιστάμενα όρια. Ε, νομίζω ότι είναι προ συμφέρον του Κοινοβουλίου να έχει μία ενιαία θέση, γιατί ε, πολύ ευκολότερα θα καταφέρουμε να πείσουμε το Συμβούλιο για τη θέση μας. Ε, ναι, ευχαριστώ. Οπότε ε, αυτό θα ψηφιστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμού και θα είμαστε έτοιμοι για την Ολομέλεια. Τώρα ερχόμαστε στα θέματα 16 και 17. Ο Ράιμερ Μπέγκε αυτή τη στιγμή είναι απασχολησμένος. αλλά ο Σούριαν έχει αναλάβει την ε, μεταφορά για το Ταμείο Αλληλεγγύης, οπότε ε, εάν πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο μας προτείνει ο Ράιμερ Μπέγκε για το Ταμείο Αλληλεγγύης στην Ιρλανδία για τη σχετική χρηματοδότηση, εάν ε, γίνεται η πρόταση να επιτραπεί αυτή η κινητοποίηση. Ε, θα ήθελα να ξέρω εάν ε, έχει λήξει η συζήτηση και αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Α, όχι, δεν θα ψηφίσουμε διότι πρέπει να περιμένουμε την τοποθέτηση του Συμβουλίου, την οποία δεν έχουμε ακόμη λάβει. Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει, τα συζητήσαμε όλα, τελειώσαμε. Οπότε τώρα προχωράμε στην ψηφοφορία, όχι όμως σχετικά με την έκθεση του Λάσλο και του Ράιμερ αλλά έχουμε να ψηφίσουμε την 2021-2022 ε, για την κινητοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και 19 και πρόκειται ε, ε, ε, κάθε φορά για μία μόνο τροπολογία την οποία ανέφερε ήδη η Μπάρμπαρα δηλαδή μία τροπολογία των Άλβαρο και Χάγκλουν ότι στις αιτήσιες εκθέσεις θα πρέπει να υπάρχει μία αξιολόγηση σχετικά με τις προσωποποιημένες ε, ε, παρεμβάσεις, δηλαδή ότι η Επιτροπή στο σημείο αυτό πρέπει να εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτού πληρώσει ποιες είναι οι επιπτώσεις του μέσου αυτού και οι δυνατότητές του για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχει αυτή η τροπολογία σε έξι εκθέσεις Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα, δηλαδή τις έξι εκθέσεις και την τροπολογία αυτή η οποία προκύπτει και στις έξι εκθέσεις αν μπορούν να ψηφιστούν on block όλα μαζί. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Μία ψήφος αρνητική, άρα εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στις μεταφορές. Στο σημείο της ημερησίας διατάξεως 25 ε, υπάρχουν πολλές μεταφορές. Λάσλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, πολλές τέτοιες μεταφορές συνδέονται με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μετά από την απόφαση που μόλις λάβαμε, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για μένα παρά μόνο να υποστηρίξω αυτές τις μεταφορές πιστώσεων. Ε, υπάρχει και μια συνολική μεταφορά μέσα στο πακέτο. Αναφέρθηκα σε αυτό με το, όταν συζητούσαμε το διορθωτικό προϋπολογισμό 10. Και... Νομίζω ότι υποστηρίζεται αυτή η συνολική μεταφορά και υπάρχουν και άλλες δύο που η μία δεν είναι στο Combo αλλά αναφέρθηκε στην αρχή και χτες νομίζω. Υπήρξε μια καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει εγγραφεί αυτό, αυτή η μεταφορά στην ημερήσια διάταξη και ρωτώ οι πολιτικές ομάδες ε, τι πιστεύουν για αυτή τη μεταφορά πιστώσης που ανέφερε ο πρόεδρος Λαμασούρ. Mm-hmm η Παριθμό 54 δηλαδή. Αφορά στις πλημμύρες στο Πακιστάν. Η Επιτροπή απέφθηνε αυτή την έκκληση προς εμάς λόγω του ανθρωπιστικού χαρακτήρα αυτής της μεταφοράς ε, και είναι και υπέρ της εικόνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να δεχτώ βέβαια ότι έχουμε κανονισμούς ε, για το χρονισμό, για τις απαιτούμενες περιόδους, για να γίνουν μεταφράσεις και το καθεξής. Τέλος πάντων, από πλευράς εισηγητού, αν υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ε, εάν δεν υπάρχει ένσταση από πλευράς των μελών της Επιτροπής μας, Πρώτα θα ήταν λογικό, κατά τη γνώμη μου, να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ψηφίσουμε. για την μεταφορά υπαριθμού 54 και αν ναι, τίθεται το ζήτημα αν ε, προτιθέμεθα να ψηφίσουμε ε, ομαδών ή όχι. Αυτά θα ήθελα να σας προτείνω, σύγητες. Μικρόφωνο. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε συνολικά όσον αφορά τις ε, μεταφορές που αναφέρονται στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή τις έξι πρώτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώσαμε. Όσο αφορά την, ε, ε, την ε, μεταφορά 54, εγώ θα είχα μία ερώτηση. Αν αυτά είναι όλα τα χρήματα τα οποία θα διαθέσει για την κατάσταση στο Αφγανιστάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι την περασμένη εβδομάδα στον τριμερή διάλογο ο Επίτροπος ανέφερε ότι στο μέλλον θα υπάρξει μία συνεδρίαση των δωρητών και η κυρία Άστον εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα διαθέσει και αυτή ε, χρήματα οπότε από ό,τι άκουσα εγώ πρόκειται για ένα πιο σημαντικό ποσό και μάλιστα ορισμένοι συνάδελφοι και εγώ ε, είπαμε ότι θα έπρεπε να μας πει πώς ε, ε, πώς προχωρά διότι η κυρία Φερέρο Βάλτνερ ερχόταν εδώ και μας ενημέρωνε για το ποσό το οποίο θα ήθελε να διαθέσει για τη βοήθεια στο Πακιστάν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ρωτώ λοιπόν αυτά είναι όλα τα χρήματα για την μεταφορά 54 ή όχι. Ας ψηφίσουμε λοιπόν πρώτα τις 6 τις, 6 μεταφορές on block και αν συμφωνείτε μετά θα προχωρήσουμε το επόμενο. Έχω μια ερώτηση προ την Επιτροπή για τι μεταφορέ που σχετίζονται με το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Προτείνει η Επιτροπή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να συνεχίσουμε να παίρνουμε κεφάλαια από το ΣΥΠΑ, από το πλαίσιο δηλαδή για τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το έχουμε κατακρίνει αυτό στο παρελθόν, έχουμε υποβάλει ερωτήσει και δημιουργούνται καταστάσει όπω η τωρινή τώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή κανονικά αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε ε, να υλοποιείται σωστά, να υπάρχουν σωστέ δαπάνε. Δεν συμβαίνει όμω αυτό, γιατί διαρκώ παίρνουμε κονδύλια από αυτό το πρόγραμμα και τα χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούμε στο Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Κάποιε επιπρόσθετε εξηγήσει μπορεί να μα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για, αυτό το, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η υποαπορρόφηση των κονδυλίων ε, του προγράμματο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr... Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα να ζητήσω από την Πρίσα να μας ενημερώσει και να μας πει αν αυτή είναι όλη η βοήθεια για το Πακιστάν. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω πρώτα στο θέμα του κυρίου Φέρμ για την πηγή των πληρωμών που γίνονται από το Ταμείο Προσαρμογής. Για τις πληρωμές λοιπόν έχουν εξηγηθεί οι λόγοι των μεταφορών ότι οι θέσεις που στοχεύουν σε παρακινδυνευμένα κεφάλαια και σε εργαλεία εγγύησης αφορούν αιτήματα που υποβάλλουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι προβλεπόμενες πιστώσεις έχουν πλήρως χρησιμοποιηθεί διότι η αποζημίωση η πραγματική πληρωμή χρειάζεται κάποιο χρόνο ανάλογα με το αν είναι εγγύηση ή παρακινδυνευμένο κεφάλαιο. Τρία με 13 χρόνια παίρνουν αυτές οι επενδύσεις και οι επιστροφές λοιπόν έρχονται με κάποια καθυστέρηση. Τα πρώτα χρόνια των προγραμμάτων το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων λέει ο ομιλητής προβλέπει ότι η Κομισιόν έχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα κονδύλια ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς πρόβλημα. Περισσότερες πληροφορίες ως προς το πόσα ακριβώς, ποια ακριβώς είναι τα ποσά σε αυτά τα trusted accounts, στα καταπιστευμένα, αυτά τα έχουμε στείλει σε ένα σημείωμα απαντητικό σε ερώτηση του κυρίου Χάγκλουντ. Και το στείλαμε στη γραμματεία σας, ίσως να έπρεπε να το διανύμει στα μέλη, διότι οι εξηγήσει που δίνονται εκεί και οι αριθμοί αναφέρονται λεπτομερώς. Τελικά βέβαια το θέμα είναι ότι η χρήση αυτών των πληρωμών για τις δύο αυτές θέσεις δεν θέτει καθόλου σε κίνδυνο τη χρήση του ταμείου διότι οι πληρωμές που απαιτούνται για να υπάρξει, για να δημιουργηθεί η νομική υποχρέωση και οι επιστροφές εξαρτώνται και από τα αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τα δε παρακινδυνευμένα σχετίζονται και με την οικονομική κατάσταση που ισχύει στη χώρα του ετούντο. του ετούντος. Ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας, τον κύκλο και τα προσαρμόζουμε αναλόγως. Ε, το δεύτερο ερώτημα για το Πακιστάν. Το αίτημα κινητοποίησης ε, της ε, βοήθειας, επίγουσας βοήθειας για το Πακιστάν έχει υποβληθεί, οι ανάγκες είναι τεράστιες και το αίτημα ζητάει να χρησιμοποιήσουμε το τελευταίο διαθέσιμο ποσό σε αυτό το απόθεμα για κατεπίγουσα βοήθεια. Αυτόν το μήνα θα το συζητήσουμε εσωτερικά και ούτως ή άλλως οτιδήποτε αποφασίσει η Κομισιόν θα βασίζεται σε αυτά που υπάρχουν στα διαθέσιμα ποσά και σε αυτά που έχουν προγραμματιστεί από το κεφάλαιο 4, ως τον τίτλο 4 μάλλον. Ένα μέρος τους έχει ήδη προγραμματιστεί για το Πακιστάν. Υπάρχουν και άλλα κονδύλια ή εργαλεία ή μέσα που μπορεί να χρειαστούν για να κανονιστούν όλα αυτά οι προτεραιότητες μεταξύ των μέσων δηλαδή για την αντιμετώπιση εκτάκτων κρίσεων και γι' αυτό σε αυτή τη φάση θα έλεγα μόνο ότι η Κομισιόν θα σας αναφέρει εν καιρό το δέοντι και εν ευθέτω χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Μέσω του υπευθύνου Αντιπροέδρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει τελειώσει το Σύριαλ αυτό. Λοιπόν, κατόπιν των εξηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να ψηφίσουμε ο μπλοκ τις έξι πρώτες μεταφορές υπέρ. Ωραία. Οπότε πάμε εις την ε, ε, μεταφορά 38. 38. Δηλαδή 29, 30, 31, 32, 33 και 34 τα ψηφίσαμε ήδη. Τώρα σχετικά με την 58. 38, 38 με συγχωρείτε. Λοιπόν, 53. Η 53 όπως είπαμε θα μεταφερθεί προς ε, ψηφοφορία είτε σήμερα το απόγευμα ή στην επόμενη συνεδρίαση. Εντάξει, θα το συζητήσουμε το απόγευμα. Αλλά πιστεύω ότι η αποδέσμευση της τροπολογίας 10 και αυτής της μεταφοράς, η μεταφορά αυτή δεν θα πάει στην Ολομέλεια, οπότε... Το ερώτημα είναι αν θα περιμένουμε για το Πακιστάν ή όχι. Τώρα η 54 και με τις εξηγήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε ήδη να δηλώσουμε ότι είμαστε υπέρ αυτής της ε, μεταφοράς. Ε Κυρία Πρόεδρε, επειδή όλοι δεν έχουν ίσως διαβάσει τα μηνύματα τα ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με αυτό. Θα, πρέπει να θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε για σήμερα το απόγευμα τη συζήτηση του εάν θα ψηφίσουμε ή όχι για να μπορέσουν οι συντονιστές να επισέλθουν στις λεπτομέρειες και να αποφασίσουν. Ναι, αλλά εγώ είμαι υπέρ του να κάνει κανείς ό,τι μπορεί όσο μπορεί πιο γρήγορα διότι οι συντονιστές λένε ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Οπότε εφόσον αυτοί συνενούν γιατί να περιμένουμε. Ας ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ της ε, μεταφοράς πιστώσεων 54, παρακαλώ σηκώσει το χέρι του. Ωραία, κατά. Κανείς. Όχι, με συγχωρείτε, ένας. Ε, ποιοι απέχουν. Κανείς. Λοιπόν, με μία αρνητική ψήφο ε, εγκρίνεται. Και 56 είναι η μεταφορά πίστοσης, πιστώσεων 56, η οποία πρέπει τώρα να ψηφιστεί. Σε αυτή τη ε, μεταφορά Ε, έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι πιστώσεις και γι' αυτό πρέπει να αυξηθεί η γραμμή. Για μένα είναι πιο σημαντικό να έχουμε ε, καλές μεταφορές και όχι καλές στατιστικές, οπότε ε, ακολουθώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εγώ πιστεύω ότι 1,7 εκατομμύρια για την Επιτροπή Μεταφορών δεν πρέπει πρέπει να το αμφισβητήσουμε αλλά αφού είμαστε υπέρ της ε, αποδοχής ποιος είναι υπέρ της αποδοχής ευχαριστώ κατά ουδής αποχές επίσης κανείς οπότε έχουμε ε, ολοκληρώσει και την μεταφορά αυτή Έχουμε χρόνο, μπορούμε παρακαλώ να επανέλθουμε εις ε, τις πλημμύρες στην Ιρλανδία διότι διάβασα πιο συγκεκριμένα ότι αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί ήδη στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου, άρα πρέπει να το διεκπαιρεώσουμε. Μπορούμε λοιπόν να το ψηφίσουμε τώρα, ακόμη και αν το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να μας δώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο. Οπότε εμείς θα έχουμε κάνει τη δουλειά μας και το Συμβούλιο θα χρειαστεί να καλύψει το, την καθυστέρηση. Λοιπόν, τότε ψηφίζουμε την έκθεση παριθμών 17 του Ράιμερ για την Ιρλανδία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κανείς. Αποχές. Κανείς. Άρα ομόφωνα εγκρίθηκε. και ο σχετικός τροποποιητικός προϋπολογισμός κατά τον Λάζλο πρέπει να υπερψηφιστεί. Ποιο συμφωνεί ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτόν τον προπολογισμό. Κατά. Κανείς. Αποχές. Πάλι κανείς. Οπότε νομίζω ότι τελειώσαμε τις δουλειές μας για σήμερα το πρωί ή όχι. Καταρχήν ναι. Πρέπει να ρωτήσουμε όμως τους σοσιαλιστές. Λοιπόν, ε, ε, ε, μου ανέθεσαν να ρωτήσω τους σοσιαλδημοκράτες τι θα κάνουν με τις μεταφορές για τις άλλες πολιτικές ομάδες, για τα λοιπά τμήματα. Ο Ντέρεκ είναι εδώ, ακόμη και αν δεν είναι ο Βλαντιμίρ Μάνκα, οπότε ο Ντέρεκ μπορεί να μας καθοδηγήσει σχετικά με τον προϋπολογισμό για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Μόλις μου λέγουν ότι οι δύο μεταφορές πιστώσεων του Κοινοβουλίου θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέλε και μετά θα αποφασίσουμε. Όλες όμως οι άλλες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν τώρα και ο Ντέρεκ έχει το λόγο. Ε, Νόμιζα ότι θα ασχολιόμαστε με το C10 και C11 τις δύο μεταφορές που όμως είχαν προβλέψει να συζητηθούν σήμερα το απόγευμα, έτσι δεν είναι. Und die anderen? Με τις υπόλοιπες ε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπόλοιπες μεταφορές. Justice up. Πρώτα θα ψηφίσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την υπαριθμόν 5. Υπέρ όλοι. Κανείς ε, κατά ούτε ε, αποχές Τώρα συζητάμε την ε, υπαριθμόν 6 για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά αποχές κανείς. Ερχόμαστε στην Επιτροπή Περιφερειών που είναι σχετικά μία πληροφόρηση. Ποιος είναι για την Info 2 του 2010 υπέρ κατά αποχές μετά Επιτροπή Περιφερειών Info υπαριθμών 3 ε, του 2010 ε, πρόκειται για 15.000 ευρώ υπέρ κατά αποχές αποφασίστηκε. Για το τρίτο και τελευταίο θέμα των, της Επιτροπής Περιφερειών, Info 4, 83.000 ευρώ, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, ωραία. Και αυτό διεκπαιρεώθηκε. Τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Οπότε, κάναμε όλες μας τις δουλειές μέχρι τις 3 το απόγευμα, οπότε θα ξαναβρεθούμε και μέχρι τότε σας χαιρετώ.